Teste 1, 2, teste. Teste 1, 2, teste. Teste 1, 2, teste.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 1, 2, 3. So please take your seats. Καθίστε παρακαλώ. So will Δύο λόγια στα γαλλικά λέει ο πρόεδρος για το ξεκίνημα. Σα εύχομαι από πλευράς τη Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημοσίας Υγείας και διατροφική Ασφάλειας και Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, υποψήφιε επίτροπε, με το χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντος και του ωκεανού ή των ωκεανών. Είναι κοινή αυτή η ακρόαση, κοινή Επιτροπής Αλίας και Επιτροπής Περιβάλλοντος. Γιατί βεβαίω αυτά τα θέματά σας είναι κοινά, κοινού ενδιαφέροντος των δύο επιτροπών μας. Όταν ε, δημοσιοποιήθηκε ο κατάλογος των υπουργικων επιτροπων Επιτρόπων, πρώτα-πρώτα αναδύθηκε η ηλικία σας κύριε υποψήφιε και είπαμε 28χρονος υποψήφιος επίτροπος. Μα μήπως είναι πρόβλημα. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Το αντίθετο πιστεύω. Ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερους 28χρονους επιτρόπους γιατί χρειαζόμαστε όλες οι γενιές και ηλικίες να είναι παρούσες στην Επιτροπή και έχετε ευξημένες ευθύνες. Σήμερα θα απαντήσετε στα ερωτήματα των βουλευτών των δύο επιτροπών. για τα θέματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος συγκεκριμένα. Ξέρουμε ότι έχετε την αρμοδιότητα και την φιλοδοξία της μηδενικής μόλυνσης για την βιοπικιλότητα, για την κυκλική οικονομία και βεβαίως όσον αφορά τον ωκεανό που είναι θέμα της Επιτροπής ε, Αλίας. Πάρα πολύ αυξημένες είναι οι ευθύνες όσον αφορά τον Green Deal, το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι η κορυφαία προτεραιότητα αυτής της νέας Επιτροπής. Οπότε προσδοκούμε συγκεκριμένε απαντήσεις σε συγκεκριμένε ερωτήσει που θα σας υποβληθούν. Και τώρα, θα δώσω τη σκητάλη στον Chris Davis. Για να σας πει πώς θα οργανωθεί η ακρόαση. Thank you. I feel obliged not to give my age. Όχι, εγώ δεν θα σας πω την ηλικία μου αντίθετα. Γιατί εδώ στο Προεδρείο φαίνεται ότι είμαι ο γυρεότερος, τέλος πάντων. Καλώς ορίσατε κύριε υποψήφιο επίτροπε, κύριε Σινκεβίτσιους. Καταλαβαίνετε ότι τα λιθουανικά μου δεν είναι τόσο δυνατά, εξού και η προφορά μου, οπότε... Α Ε, βέβαια, εσεί αντίθετα ε, ε, περάσατε τρία χρόνια στην Ουαλία στο Πανεπιστήμιο. Για να αρχίσουμε τώρα το πώ θα ε, συζητήσουμε. Ξεκινούμε από την ανακτήρια αρχή σα δήλωση, 15 λεπτά και κατόπιν θα δοθεί ο λόγο στου συμβουλευτέ του επιτροπών, 25 δηλαδή, ε, για την πρώτη ερώτηση έχουν μισό λεπτό οι συνάδελφοι. Οπότε ε, θα ήθελα να του παρακαλέσω όμω να μην χρησιμοποιήσουν όλα τα 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο ψήφιο επίτροπο θα έχει δύο λεπτά για να σα απαντήσει και ο ερωτή σα θα έχει επερώτηση ανάλογα με το πόσο χρόνο έχει, του έχει ε, περισσέψει την πρώτη ε, ερώτηση και θα απαντήσει σε ένα λεπτό στην επερώτηση ο κύριος Υπουργός Οπότε έχουμε τον ε, πρώτο γύρο των ερωταπαντήσεων για περιβαλλοντικά θέματα, ο πρώτος γύρος και ο δεύτερος για θέματα αλληλείας. Στο τέλος. Θα έχει ένα πεντάλεπτο για την καταληκτική τελική του δήλωση ο υποψήφιος επίτροπος. Και μου λένε να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σε όλες τις γλώσσες διερμηνία. Μπορείτε όλοι να μιλήσετε τη μητρική σα γλώσσα. Παρακαλώ, μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα γιατί οι διερμηνεί δεν θα προφτάσουν να σα ε, μεταφράσουν. Μεταδίδεται στο ίντερνετ αυτή μας η συνεδρίαση και μπορεί κανείς να δει και το βίντεο γιατί θα υπάρξει ε, βιντεοσκόπηση της ε, ανάκρισης. Έχετε κύριε Πίτροπε την, ε, το χαρτοφυλάκιο σα αυτό, δηλαδή θα πρέπει δηλαδή να πετύχει τη βιωσιμότητα όσο γίνεται περισσότερο, να σταματήσει η υπεραλίευση και όλα αυτά μέχρι το τέλο τη επόμενη χρονιά. να εξασφαλίσετε επίση το τι θα γίνει με τι ε, εκφορτώσει, να τηρηθούν οι απαγορεύσει σχετικέ που δεν ε, τηρούνται, θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται διάφορε ουσίε, βλαπτικέ για το περιβάλλον και έτσι να μην έχουμε και από αυτό το υπεραλίευση, επομένω τίποτα, λίγα πράγματα, ψηλό πράγματα. Καλά, καλά, μετά θα τα πούμε μετά για την Ιταλία. Χαλαρώστε πρώτα-πρώτα περιβάλλον. Έχετε το λόγο. Audible members, good afternoon. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλησπέρα και σα ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση αυτή για να σας αναπτύξω το όραμά μου για την επόμενη θητεία. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ ως ο πρώτος υποψήφιος επίτροπο που γεννήθηκε μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Είναι ένα σημάδι εμπιστοσύνη στη γενιά μου. Μια γενιά με ένα ευρωπαϊκό ιδεώδες στο DNA της. Για εμένα η Ευρώπη σημαίνει ελευθερία, ευκαιρία και ανοιχτή ορίζοντες. Ταυτόχρονα σημαίνει και ανάληψη ευθύνης. Το τελευταίο κύμα αυτό των κλιματικών απερκειών δείχνει πως οι επόμενες γενιές είναι έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ως ε, μέρος και εγώ της ε, νέας γενιάς είμαι αποφασισμένος να αναλάβω την σκητάλη. Για εμάς το 2050 δεν είναι ένας στόχος σε ένα κομμάτι χαρτί, θα το ζήσουμε. Τώρα θα μιλήσω την μητρική μου. Ε, η πολιτική μου σταδιοδρομία ξεκίνησε με τις εκλογές ε, στο Βίλνιους, έγινα βουλευτής ε, και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Τα τελευταία χρόνια ήμουν υπουργό των Οικονομικών και έτσι έχω μάθει να υπηρετώ τους συμπολίτες μου, να αντιλαμβάνομαι τα προβλήματά τους όπως ε, το κάνετε και εσείς ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη χώρα μου για την ευκαιρία που μου έδωσε να έχω αυτήν την σταδιοδρομία. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, της ψηφιακής οικονομίας και της βιομηχανίας, της καινοτομίας και του κοινωνικού πλούτου δεν είναι αντιφατικά αυτά. Οι προκλήσεις είναι και ευκαιρίες και οδηγούν σε μια κοινωνία με μεγαλύτερη ευμερία. Το ταξίδι μας προς έναν πράσινο πλανήτη με μηδενικές εκπομπές έχει ξεκινήσει. Θα είναι δύσκολο. Ως Επίτροπος θα κάνω οτιδήποτε είναι δυνατόν για να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Είμαστε πολλοί σε αυτήν την πορεία. Το βλέπουμε αυτό από τις διαμαρτυρίες για το κλίμα, τις ε, ευρωεκλογέ και το ευρωβαρόμετρο. 92% των Ευρωπαίων θέλουν μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Πρέπει να ακούσουμε λοιπόν. Και παρουσιάζοντα ε, το Green New Deal, ε, η πρόεδρο Φόντερ Λάιν έχει κάνει ακριβώ αυτό. Η μεγαλύτερη μου φιλοδοξία, αν με ορίσετε, θα είναι να γίνει το πράσινο New Deal πραγματικότητα και να λειτουργήσει για τους ωκεανούς, για το περιβάλλον και για τους πολίτες μας. Πρέπει να είμαστε στο επίκεντρο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ίσως προξένησε έκπληξη κάποιους το ότι υπάρχουν οι ωκεανοί στο όνομα του χαρτοφυλακίου μου και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας ε, γιατί θέλετε μια διαβεβαίωση ότι θα ασχολείται και με τους ψαράδες ο νέος επίτροπος. Σας διαβεβαιώ λοιπόν τώρα. Ζούμε σε έναν γαλάζιο πλανήτη. Τα αλληλευτικά αλλιεύματα, τα αλληλευτικά με συγχωρείτε από θέματα και οι ωκεανοί πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο τη πολιτική μα. Ναι, αλληλεία αλλά και περιβάλλον. Πρέπει να δούμε και την κλιματική αλλαγή. Όπω είδαμε από την τελευταία έκθεση τη διακυβερνητική διάσκεψη, έχουμε ρήπανση πλέον σε ολόκληρη την ε, διατροφική αλυσίδα. Έχουμε τα αζωτούχα από τα λιπάσματα, τα οποία προκαλούνται κρέζο στην ε, θάλασσα. Οι υγιεί ε, ωκεανοί σημαίνουν ε, υγιή αλλιεύματα και αυτό σημαίνει υγιείς κοινότητε, ψαράδων και βεβαίως ε, και υγιείς πολίτες με λιγότερες αρρώστιε. Πάντα εγώ προσπαθώ λοιπόν να συνεργάζομαι και το ίδιο θα κάνω και στην θητεία μου, θα συνεργάζομαι μαζί σας. Υπάρχουν λοιπόν τρία βασικά στοιχεία στο ευρωπαϊκό πράσινο New Deal. Αυτό θα γίνει υπό την ηγεσία του Φραντ Τίμερμανς, ο οποίος βεβαίω ως πιο έμπειρος θα με καθοδηγήσει. Οι τομεί αυτοί είναι η βιοπικιλότητα, η κυκλική οικονομία και η μηδενική ρήπανση. Η βιοπικιλότητα εξαφανίζεται. Η έκτη μεγάλη εξαφάνιση των ειδών έχει ήδη ξεκινήσει. Εάν με ορίσετε λοιπόν αρμόδιο θα εκπροσωπήσω την Ευρώπη στην σχετική σύνοδο στην Κίνα το επόμενο έτος. Έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την πορεία αυτή. Θα ήθελα να επιστρέψω λοιπόν με τρία πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι ανάλογο με τους στόχους του Παρισίου για την βιοπικιλότητα. Δεύτερον, θεωρώ ότι οι εθνικές δεσμεύσεις για την επίτευξη των ε, στόχων θα μας βοηθήσουν να το επιτύχουμε. Τρίτον, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό για να μετράμε την πρόοδο. Οι εταίροι μα αναζητούν και θέλουν από εμά αυξημένη στήριξη για να πολεμήσουμε την απώλεια τη βιοπικιλότητα. αλλά η διεθνή μα αξιοπιστία εξαρτάται και από την πρόοδο στο ιστορικό. Υγείστε δια του παραδείγματο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα σημεία τα οποία εφίστανται πίεση, τα δάση, τα εδάφη και βεβαίως το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε λύσεις από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Η νέα πρόεδρος απαιτεί νέες προδιαγραφές για την βιοπικιλότητα στο εμπόριο, στην βιομηχανία, στη γεωργία και στην οικονομία. Και είμαι αποφασισμένος να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Αλλά και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Στο να ενταχθεί η βιοπικιλότητα σε όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η δεύτερη μου προτεραιότητα θα είναι η κυκλική οικονομία. Θέλω να έρθει στο προσκήνιο, να μην είναι απλά κούφια λόγια. Εάν αυξηθεί η κυκλική οικονομία τεσσάρων υλικών, του χάλιβα, του τσιμέντου, του αλουμινίου και των πλαστικών, θα μειώσουμε τις εκπομπές μας στο μισό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τρεις βασικές δέσμες δράσης εδώ πέρα θα μπορούσαμε να δούμε τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης με οικολογικό σχεδιασμό. Επίσης θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την κυκλικότητα σε νέους τομείς όπως τα υφάσματα, οι κατασκευές, τα τρόφιμα και ο τομέας πληροφορικής. Η δεύτερη δέσμη είναι να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι όταν κάνουν επιλογές. Όταν βλέπουν ένα προϊόν που λέει ότι είναι πράσινο θα πρέπει να το πιστεύουν. Και τρίτο πρέπει να πάμε πέρα από την ανακύκλωση. Δεν θέλουμε απλά να μειώσουμε τα απόβλητα, θέλουμε να μην δημιουργούνται καν. Όπου είναι αυτό δυνατόν, στι κατασκευέ, στα υφάσματα και σε πολλού άλλου τομεί. Η τελευταία μου δράση θα είναι η μηδενική ρήπανση. Ω πατέρα, ω πολίτη και ω Ευρωπαίο Επίτροπο θέλω η ρήπανση να ανοίξει στο παρελθόν. Θέλω μια Ευρώπη με καθαρό αέρα, καθαρό νερό, και μηδενική ρήπανση. Αυτό θα απαιτήσει μια νέα προσέγγιση, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες. Για τις χημικές ουσίες θα πρέπει να δούμε τις επικίνδυνες από αυτές και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Για το νερό. Αυτό θα σημαίνει να δούμε τα μικροπλαστικά, τις διατροφικές ουσίες και τις φαρμακευτικές ουσίες στο νερό και θα πρέπει να έχουμε μια νέα προσέγγιση στα ζυζανιοκτώνα σε συνεργασία με την Επίτροπο για την Υγεία σε μια στρατηγική από το χωράφι μέχρι το πιάτο για να μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικέ στα χημικά φάρμακα. Πάντα με βάση την επιστήμη. Ε, κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να συνεχιστεί και στο 8 πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον, για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Τώρα θα αναφερθώ στους στόχους μου για τους ωκεανούς. Ο πρώτος είναι η πλήρης εφαρμογή Τη πολιτική αλληλεία. Πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία. Όταν η αλληλεία είναι βιώσιμη, τα κέρδη αυξάνονται. Το 2022 θα αξιολογήσω την πολιτική αλληλεία για να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώ. Χρειαζόμαστε μια πολιτική η οποία θα λειτουργεί για του αλληλεί, για τι παράκτητε κοινότητε και για το περιβάλλον. Βεβαίω έχουμε και πολλέ διαφορέ Αυτό το οποίο ισχύει στην Βόρεια Θάλασσα μπορεί να μην λειτουργεί στη Μεσόγειο κάθε θάλασσα είναι διαφορετική και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Οι προσπάθειε μας για, υγιούς, για υγιείς παραγωγικούς ε, δεν μπορούν να σταματάνε στα σύνορά μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να επιβάλλω τις αρχές της ε, βιωσιμότητα παγκοσμίω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και στους ωκεανούς. Θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν για να απαγορευτούν ορισμένες βλάπτικες τεχνικές αλληλεία και για αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτων. Σε διεθνή υδάτα, όπως ε, η Ανταρκτική, που είναι ακόμα ανέγκυχτα, χρειάζονται νέοι κανόνες για την στήριξη της ε, βιοπικιλότητα. Και θα συνεχίσω την ε, μάχη μα κατά τη ε, η λαθραλία απειλεί τους υπεύθυνου ψαράδες, ειδικά μικρής κλίμακας, που υφίστανται άγριο ανταγωνισμό και βλέπουν τους πόρους να μειώνονται. Το ψάριμα είναι ένα ευγενές επάγγελμα. Κάθε μέρα οι ψαράδες εργάζονται σκληρά για να μας δίνουν πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας. Πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους. Η ευημερία των παραθαλάσσιων ε, κοινοτήτων κινδυνεύει. Η πολιτική μας κατά της λαθραλίας θεωρείται καλύτερη στον κόσμο, αλλά βέβαια οι κανόνες δεν έχουν κανένα νόημα χωρίς εφαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να διασφαλίζει ίσους ανταγωνισμού. Θα αντιμετωπίσω τις ελλείψεις όπου τις βρω και τρίτον θέλω να επενδύσουμε στα αηφόρα θαλασσινά. Τα ψάρια και τα θαλασσινά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε 5.000 ε, τόνους ε, ψάρια και 4,1 εκατομμύρια τόνους ε, από τις ηχθειοκαλλιέργειες. Έχουμε λοιπόν την γαλάζια οικονομία όπως τη λέμε, το οποίο αφορά από την θαλάσσια χωροταξία, τις ΑΠΕ στην θάλασσα, τις επενδύσεις στη θάλασσα. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι συνολικά εργάζονται στην θαλάσσια οικονομία. Μπορεί να ακούγεται μικρό αριθμό. Για εμένα είναι μεγαλύτερο από τον πληθυσμό τη χώρα μου. Όπως με υπενθύμησε και η πρόεδρος, η νομοθεσία είναι μόνο τόσο καλή όσο η εφαρμογή τη. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η εφαρμογή σε όλου του τομεί τη πολιτική, χρησιμοποιώντα κάθε μέσο που έχω στην διάθεσή μου. Τον διάλογο, την έκθεση εφαρμογής νομοθεσίας, διαδικασίες επί παραβάση. Χρειαζόμαστε λοιπόν νόμους οι οποίοι θα λειτουργούν για τους πολίτες, για το περιβάλλον και για τους ωκεανούς και τα ψάρια και τις επιχειρήσεις. Κυρίε και κύριοι, αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Η επιτυχία μας εξαρτάται από την συνεργασία. Θα με βλέπετε λοιπόν τακτικά στους διαδρόμους, στις συνεδριάσεις σας. Θα είμαι εδώ πέρα για συζήτηση μαζί σας, για διμερείς συναντήσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες άμεσες επαφές. Θα πάω στις χώρες σας, όχι μόνο στις πρωτεύουσε, αλλά και στις περιφέρειες και στις παράκτιες κοινότητε. Και σας ευχαριστώ για τις προσκλήσεις που έχω ήδη λάβει. Όπως είπα στην αρχή, πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες. Εσείς είστε οι αιρετοί εκπρόσωποι τους. Και σας εμπιστεύονται. Χαίρομαι λοιπόν που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια και τώρα είμαι στην διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ε, με τις πρώτες επτά ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΙΟΥ πολιτικές ομάδες και έπειτα θα ακούσουμε επτά από την Επιτροπή Αλίας. Ξεκινούμε λοιπόν με το ΕΛΚΑ και την Τζέσικα Πολφιαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Ριστέντα Επίτροπε. Θα μιλήσω σου ειδικά. τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά είναι πολύ σημαντικά για τον πλανήτη. Έχουμε κοινού στόχους, αλλά για να τους πετύχουμε πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην έρευνα. Η έρευνα τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα δάση δεν δραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και αν τα διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση θα μπορούν να συγκρατούν το διοξίδιο του άνθρακα. Άρα τα δάση βοηθούν την προστασία του περιβάλλοντος. Βοηθούν επίσης ε, όχι μόνο για να μας παρέχουν θέρμες, αλλά και για να επιβιώνουμε. Η δασοκομεία λοιπόν είναι προτεραιότητα. Επίσης, ε, στα δάση είναι πολύ μεγάλη βιοπικιλότητα. Η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα κάνει λόγο για τα δάση, πολύ συγκεκριμένα. Το σημαντικό είναι να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης δασοκομείας και της προστασίας της βιοπικιλότητας. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι καύσονες, οι ξηρασίες των τελευταίων ετών έπληξαν ε, τα δάση ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ζώα που κατοικούν στα δάση έχουν υποφέρει πολύ από αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν περισσότερο από ποτέ σήμερα να προστατεύσουμε τα δάση. Υπάρχουν και τρία εκατομμύρια άνθρωποι που απασχολούνται στον τομέα αυτό. Η δασοκομεία πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, περιβαλλοντικές δυσκολίες. Εσείς λοιπόν ως επίτροπος, αν οριστείτε, πώς θα φροντίσετε να ληφθούν ε, δεόντως υπόψη στη μελλοντική στρατηγική προστασία της βιοπικιλότητας ε, όσα προσφέρουν τα δάση. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, μην ξεπερνάτε το 1,5 λεπτό και έχετε 30 δεύτερα για επερώτηση. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. Απάντηση. Okay. Thank you. Uh, thank you for your question. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ξέρω ότι έχετε ζητήσει να γίνουν μέτρα, να ληφθούν μέτρα κατά της αποψήλωση των δασών. Σίγουρα είναι σημαντικά τα δάση, το 40% της ε, έκτασης, επιφάνειας της καλύπτεται από δάση, τα οποία πρέπει να τα προστατεύουμε και να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Βέβαια, σημαντικό είναι να λάβουμε είναι και τις νέες ε, προκλήσεις οι χώρες μέλη λοιπόν πρέπει να έχουν αποτελεσματικά ε, σχέδια διαχείρισης ε, των δασών λόγω των δασικών πυρκαγιών. Είδαμε τι έγινε στον Αμαζόνιο, στη Σιβηρία. Αλλά και στην Ελλάδα τα ίδια γίνονται κάθε χρόνο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνούμε τα διαχειριστικά σχέδια. Επίσης, δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα ε, η νομοθεσία για την ξυλία σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει λοιπόν ομοιομορφία μεταξύ των κρατών μελών. Βέβαια, ο ακρογωνιαίο λίθο προστασία των δασών είναι σίγουρα η στρατηγική για την βιοπικιλότητα. Η στρατηγική αυτή είναι ένα από του βασικού πυλώνε και τη νέα πράσινη ε, συμφωνία. γιατί κατ' εμέ, αν δεν έχουμε αποτελεσματική διαχείριση τη βιοπικιλότητας, δεν θα έχουμε και μια αποτελεσματική πράσινη συμφωνία. Άρα πρέπει ε, την υποβάθμιση των δασών, ε, την διατήρηση να τα έχουμε προτεραιότητα και τις προτεραιότητες, ε, τις περιοχές Natura 2000 να τις έχουμε σε προτεραιότητα. Δεν μιλάω μόνο για τις ε, προστατευόμενες αυτές περιοχές, μπορεί να είναι 25, 30, 35%. Μιλάω για πραγματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τις περιοχές αυτές. Δεν λέω να μην γίνεται καμιά ανθρώπινη δραστηριότητα εκεί, αλλά ε, να γίνεται με μέτρο ότι γίνεται και να υπάρχει έλεγχος. Θέλουμε συγκεκριμένες ενέργειες και βέβαια πάνω απ' όλα θέλουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση. 30 δευτερόλεπτα για την ε, ερώτηση. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα συνεργαστείτε και με άλλους επιτρόπους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε με τον Φραν Τίμερμα συγκεκριμένα πώς θα συνεργαστείτε και πώς θα επιμείνετε ώστε να λαμβάνετε υπόψη το δυναμικό των δασών σε όλες τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Απάντηση. Πολύ καλό ερώτημα και νομίζω αυτό είναι και το κλειδί της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε από κοινού με τον κύριο Φραν Τίμερμανς. Στο δικό μου το, στην δική μου την επιστολή που έχω την εντολή μου, αναφέρεται σαφώς η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα και φυσικά και θα πρέπει να συνεργαστώ με τον κύριο Τίμερμαν, ώστε να λαμβάνετε υπόψη την επιτυχία αυτή στη γεωργία, στην ενέργεια, στις μεταφορές και σε άλλες δηλαδή πολιτικές. Οτιδήποτε προξενεί σήμερα προβλήματα. Τον αφανισμό ειδών, χλωρίδας και πανίδας. Αυτά πρέπει να δούμε. Και ε, σας το λέω κατηγορηματικά. Επειδή τα συζητούμε αυτά, λέμε ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι, περισσότερα χρήματα. Το σημαντικό όμως είναι να είναι στρατηγική η στόχη αυτή. Διότι υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, οι οποίοι έχουν να κάνουν τη βιοπικιλότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα βλέπουμε απομονωμένα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι τώρα ό,τι κάναμε στη Γεωργία και να έχουμε πιο βιώσιμους στόχους για τη βιοπικιλότητα 2030. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Θέσαρ Λουένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να καταρρύψετε το τείχος του αρνητισμού και της ε, αδιαφορίας ε, και έχουμε πάρα πολλούς πρόορους θανάτους, ε, χρόνιες ασθένειες, τεράστιο κόστος για τα συστήματα υγείας η περιβαλλοντική ρήπανση μπορεί να σώσει ζωές και να μειώσει και τις ασθένειες. Ε, λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε για να μειωθούν οι εκπομπές από τις βιομηχανίες, ε, μεταφορές, ε, από τα σπίτια κτλ. Και πώς θα τηρούν όλα τα κράτη-μέλη τα πρότυπα για την προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. Θα λάβετε υπόψη ε, τις ε, τελευταίες προτάσεις ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Υγείας και θα προτείνετε πιο αυστηρά πρότυπα για τις εκπομπές από τα οχήματα αεροσύντη. Please go Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Πραγματικά δεν είναι καθόλου λογικό να πεθαίνουν λόγω ατμοσφαιρικής ρήπας 300.000 άνθρωποι το χρόνο και η οικονομία είναι 24 δις το χρόνο. Δηλαδή απόλυες υπάρχουν και τις βλέπουμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει τους νόμους που έχουμε θεσπίσει να τους εφαρμόζουμε πλήρως. Και σε ό,τι αφορά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, για τα σωματίδια τα αιωρούμενα για παράδειγμα έχουμε συμπεριλάβει ε, τις διατάξεις αυτές στην νομοθεσία μας ήδη από το 2006. Θέλουμε λοιπόν ξεκάθαρα σχέδια δράσης. Πρώτον, μηδενική ανοχή ε, σε περίπτωση μη συμμόρφωση ε, με τα πρότυπα για την ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Φυσικά θα πρέπει να δούμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, χαρτογράφηση, προσαρμογή στι συστάσει Παγκοσμίου υγείας Υγεία και βεβαίω για τις πόλεις διάλογος και μηχανισμοί. Αυτό είναι η προτεραιότητα για να προσαρμοστούν οι πόλεις και οι χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά ενδεχόμενε καθαρέ περιοχέ, ποιε αρχέ μπορεί να επιβάλλουν περιορισμού στην κυκλοφορία ή ελεύθερε, απαλλαγμένε από διοξείδιο του άνθρακα ζώνε. Σε ό,τι αφορά το Euro 7, ε, υπάρχει μια εντολή. Ε, μέσα σε πέντε χρόνια νομίζω ότι μπορούμε να το έχουμε, το Euro 7, το Euro 7. Μαζί με τον Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά θα συνεργαστώ σε αυτό το θέμα. Για τα τζελοκίνητα οχήματα που ρηπαίνουν, όπω και ο Επίτροπο Ιστορική Αγορά θα εφαρμόσετε την υποχρεωτική απόσυρση αυτών των οχημάτων σε όλη την επικράτηση τη Ένωση και τέλο. Ε, μαζί ε, θα προσπαθήσετε και με βάση και το Dieselgate, το σκάνδαλο που ήδη το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στην Ευρώπη, επειδή είπατε ότι γεννηθήκατε μετά την πτώση του τείχου, ε, επαναλαμβάνω, ρίξτε το τείχο τη αδιαφορία, ρίξτε το τείχο του αρνητισμού απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Απάντηση. Ναι, σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα, το Dieselgate. Μας δίδαξε ένα πολύ σκληρό μάθημα. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναυπάρξει Dieselgate. Αυτό είναι το σίγουρο. Και νομίζω το αντιλαμβάνεται και αυτοκινητοβιομηχανία όλο και περισσότερο αυτό σε ό,τι αφορά την απόσυρση οχημάτων. Ε, ακούστε, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο πλαίσιο έγκριση τύπου που θα ισχύσει από 1 Σεπτεμβρίου του 2020 και θα δοθεί αυτή η δυνατότητα επομένω. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία μα να είναι ανταγωνιστική. Και πρέπει να δούμε προ τα που οδεύει η βιομηχανία. Υδρογόνο, ρεύμα, ηλεκτροκίνηση. Θα πρέπει δηλαδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες μας που είναι κορυφαίες παγκοσμίω ε, να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Ε, μπορεί να μην καταφέρουν να είναι τόσο επιτυχημένοι σε κάποιοι Αμερικανοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά τουλάχιστον να ανακτήσουν κάπως το χαμένο έδαφος, ε, να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Και βέβαια πρέπει να προωθήσουμε τα καθαρά εναλλακτικά καύσιμα. Ευχαριστώ. Thank you. You can go to the end of your sentence. No problem. It, it would be one more sentence. Α, είχε Όχι, είχε ακόμα. Ακόμα μια φρασούλα. Καλά. Κρατήστε την για την επόμενη ερώτηση και τώρα η Φρεντερική Ρίσκ. Καλημέρα κύριε Συγκεβίτσιος. Εδώ, εδώ είμαι έχετε δύο ρεκόρ του και του πιο νέου επιτρόπου και επίσης ε, ότι έχετε το νοκιανό στο χαρτοφυλάκιο πάρα πολύ συμπατικό αυτό το θέμα είναι βέβαια αν θα τα πετύχετε όλα αυτά εγώ ξέρετε ε, για τα υλικά της αλίας και για την αλία έχω αναλάβει μια έκθεση και είναι το θέμα η ρήπανση, η μόλυνση, το πλαστικό και έχουμε αυτό το 70% οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι και στη σελίδα 11 λέτε ότι θέλω να δούμε τι μπορεί να γίνει με το πλαστικό και να έχουμε βιοδιαλυτά υλικά τα οποία να μην βλέπουν το περιβάλλον. Για πέστε μας, είναι δυνατόν σχετικά με αυτό να έχετε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ακριβώς όσον αφορά αυτή τα βιοδιαλυτά πλαστικά, τι μπορεί να γίνει. Γιατί όπως ξέρετε, σήμερα δεν υπάρχει πρότυπο ευρωπαϊκό τίποτα όσον αφορά τις πραγματικές συνθήκες για τις θάλασσες. Υπό αυτές τις συνθήκες είσαστε βέβαιοι ότι διαλέξατε τη σωστή μέθοδο. Θα πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να δοθεί μια όθηση στα πράγματα. Να μην έχετε έναν στόχο φαραωνικό που δεν αλλάζει τίποτα και είναι εις βάρος των πάντων αλλιέων και καταναλωτών. Επίσης, τι γίνεται με τις πλαστικές συσκευασίες που το θίξατε. Υπάρχει σχετική οδηγία που αν την περιμένουμε για του χρόνο εσείς θέλετε να υποσχεθείτε ότι κάτι θα γίνει και θα υπάρξει κάποια νομοθεσία με ποσοτική αποτίμηση και φυσικά δεσμευτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Επίτροπος. Ναι, συμφωνώ ότι το business as usual αν δεν αλλάξει τίποτα τότε θα καταλήξουμε σε περισσότερο πλαστικό. Περισσότερο πλαστικά από όσα ψάρια. Και χέρι-χέρι με το κοινοβούλιο, θέλω να δούμε τι θα γίνει με πλαστικά μιας χρήσεως ε, και δεν θα μπει φρένο σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε και θα επιδιώξω 100% να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική, αλλά το επόμενο βήμα θα είναι τα μικροπλαστικά. Σε κλωστοφαντουργικά, ε, σε πλάστικα και θα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο και να δούμε πώς τα βιοδιασπόμενα θα είναι φτιαγμένα με τα σωστά χημικά. Άλλο πολύ σημαντικό. Μην υπάρχει υπερβολική συσκευασία, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο. Θα πρέπει να δούμε τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις ε, και αυτοί θα πρέπει να περικόψουν. Δεν θα είμαστε βέβαια μόνοι στην προσπάθεια γιατί Διεθνώς γίνεται προσπάθεια στο G7, στον ΟΗΕ και επομένω με τις ε, διμερείς επαφές με τους εταίρους μας νομίζω ότι έχουμε κάνει πράγματα που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και θα συνεχίσουμε. Ο πρόεδρος. 15 δευτερόλεπτα για την επερώτηση. Ναι, καταλαβαίνω το ότι υπόσχεται για τα μικροπλαστικά προσπάθειες ο Επίτροπος, αλλά κάτι για την οικοσύλληψη. Ε, τι θα γίνει, θα ανακυκλώνονται αυτά τα πλαστικά, μπορείτε να βάλετε για τα μικροπλαστικά κάποια φίλτρα στα πλυντήρια, ούτω ώστε να μην καταλήγει το δηλητήριο που καταλήγει τώρα στα ποτάμια μας. Ναι, πολύ σωστά τα είπατε. Είναι ακόμα ένα πρόβλημα τα πλυντήρια και γι' αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί η χρήση του eco design. Κατά τη γνώμη μου όμως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, εδώ γεννήθηκε η ιδέα και θυμάμαι τις πρώτες συζητήσεις για το eco design. Και θυμάμαι ότι λέγανε και που θα, κατα... θα καταντήσετε να νομοθετήσετε και για τους γλόμπους. Όμως, έγινε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας όσο της Ιταλίας. Με αυτή τη διαφορά. Στην Ιταλία σε ένα χρόνο δηλαδή. Ενώ, άρα θα πρέπει ο πύχης να παραμείνει ψηλά, να σπάσει αυτός το τοξικός κύκλος και είναι σημαντικό τα πλαστικά να φτιάχνονται από χημικές ουσίες μη τοξικές και κατόπιν να ξαναμπαίνουν αυτές οι ουσίες στην κυκλική οικονομία. Και η κοινοτομία προβλέπει πολλές τέτοιες εφαρμογές. Πράσινη. Γκίγκολτ. Η υποψήφια <coughs> uh, in your written... Οι υποψήφοι ε, τονίζεται γραπτές ότι οι πιο ευπαθείς ε, στην Ευρώπη ε, επηρεάζονται δυσανάλογα από τους κινδύνους ε, για την υγεία. Και έχετε δίκιο. Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, ε, τα επίμονα χημικά και τα νανοηλικά. Σύμφωνα με τις μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο αριθμό των ανθρώπων που επηρεάζεται από ενδοκρινικές διαταχές αυξάνεται. Υπολογίζεται ότι 25% των παιδιών στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων και τα δικά μου παιδιά, υποφέρουν από τα λεγόμενα δόντια του καρχαρία, μια ασθένεια η οποία σχετίζεται με τον πισφενόλ α, ε, γνωστή ουσία η οποία διαταράσσει το ενδοκρινικό. Τι θα κάνετε λοιπόν για να προστατεύσετε τα παιδιά μας από τέτοιες ουσίες. Η λιδία λίθος θα είναι τελικά εάν θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με αυτά τα υλικά, τα νανοηλικά, το κοκτέιλ και την έκθεση στα χημικές ουσίες από προϊόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Thank you very much for your question. And I... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ερώτησή σας ε, και την αντιλαμβάνομαι όχι ως υποψήφιος ε, επιτροπός αλλά ως πατέρας, ως καταναλωτής. Έχω ένα ε, παιδί 3,5 ετών και θα γεννηθεί και η κόρη μου ε, κάποια στιγμή μες τον Οκτώβριο. Λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι. Οι χημικές ουσίες ε, μας περιβάλλουν στην καθημερινή μας ζωή και υπάρχουν πάνω από 100 ευρωπαϊκά νομοθετήματα για το θέμα. Οπότε πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί όπως αναφέρθηκε ακριβώς στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και να διασφαλίσουμε ότι τα ασφαλή τα υλικά θα είναι ασφαλή και μη τοξικά. Είμαστε πραγματικά πρώτοι στον ε, κόσμο. Νομοθεσία σαν το ρίτσι δεν υπάρχει αλλού. Οπότε πρέπει να προωθήσουμε την ε, καινοτομία. Και συγκεκριμένα για τους ε, διαταράκτες του ενδοκρινικού, οπωσδήποτε πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική που θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Το σημαντικότερο βεβαίως είναι ότι βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης και οι διαταράκτες του ενδοκρινικού πρέπει να τυποποιηθούν και να τις δούμε στο ίδιο πλαίσιο με τις ε, ουσίες CMR. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευπαθείς, ε, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, ε, να φύγουν οι ουσίες αυτές από τα καλλιντικά, ό,τι έρχεται σε επαφή με το φαγητό όλα αυτά. Αν μου επιτρέπετε, σας ευχαριστώ για αυτή τη δέσμευση. Για τη στρατηγική για το μη τοξικό περιβάλλον θα ε, έχετε αποτελέσματα και στα τέσσερα μέτωπα που ανέφερα. Κοιτάξτε, θα έχουμε τρεις πυλώνες σε αυτήν την πολιτική. Ένα σχέδιο για καθαρό νερό, για καθαρό αέρα και για ένα μη τοξικό περιβάλλον που θα πρέπει να προχωρήσει παραπέρα. Βεβαίω, έχουμε κάνει πολλά αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η δουλειά έχει γίνει αρκετά καλά. Ε, Ξαναείδαμε την ομοθεσία και τις χημικές ουσίες. Το REACH αναθεωρήθηκε. Έχουμε τους 16 στόχους, οπότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ για το ID, κυρία Μπαλτασάρη. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό το χαρτοφυλάκιο και είμαι σίγουρη ότι το έργο σας δεν θα διέπεται από δουλειά στο γόνατο, αλλά από μία λογική διαχρονική. Όμως έχουμε κάποιες επιστημονικές μελέτες με επιστημονική μέθοδο, με την κοινή λογική για τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Είμαι γιατρός και δεν ξέρω πρόκειται να κάνετε ό,τι ανακοινώσατε για τους, τις περιβαλλοντικές ανακοινώσεις και επιπτώσεις των φαρμάκων. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κατάλοιπα στα υπόγεια και στα υπέργεια ύδατα και στα ζώα. Ε, όλα αυτά είναι κακά για το περιβάλλον. Βέβαια, αυτά τα φάρμακα ίσως δεν είναι σε αρκετή συγκέντρωση για να είναι επικίνδυνα, αλλά επί τη βάση των όσων λένε οι επιστήμονες δεν θα πρέπει να εφαρμόσετε την αρχή της ε, πρόληψης. Τι θα κάνετε, η νέα Επιτροπή πρόκειται να θεσπίσει ένα νομοθέτημα για αυτό το πρόβλημα των φαρμάκων. Thank you. Uh, thank you for your question. ευχαριστώ για την ερώτησή σας, λέει ο Επίτροπος. Ήδη τα φάρμακα καλύπτονται από την νομοθεσία για τα ύδατα όσον αφορά δηλαδή τη χημική μόλυνση. Εδώ και καιρό. Είναι σημαντικό και το παρακολουθούμε και τώρα κάνουμε fitness check και στα πλαίσια της οδηγίας πλαισίου και όσον αφορά τα ποιοτικά πρότυπα των υδάτων, οπότε θα κάνουμε την αξιολόγηση και να δούμε αν χρειάζεται να αλλάξουμε το ισχύον καθεστώς και διαπιστώνουμε όλοι ότι τα φάρμακα είναι όλα ένα και πιο επικίνδυνα οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην μπαίνουν στα ύδατα. Φυσικά και χρειάζεται πρόληψη. Βεβαίως και θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια του στόχου μας για μηδενική μόλυνση και ρήπανση. In conclusione, la Περασματικά, η Επιτροπή θα θεσπίσει ήου ένα νομοθέτημα. Και τι θα κάνετε, κανονισμό ή οδηγία ποιο είναι το πιο δόκιμο, ούτω ώστε η εθνική κυριαρχία και η επικουρικότητα να γίνουν σεβαστά. Okay, thank you. Uh, thank ε, Ο Επίτροπος, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, βέβαια, εγώ είναι πρόημο να το πούμε, αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα μαζί. Ήδη τα φάρμακα από την νομοθεσία για τα υδατά, αλλά έχουμε και την οδηγία πλαίσιο που τώρα σε διαδικασία ε, μελέτης και αναθεώρησης, οπότε και θα δούμε εάν τελικά θα προσθέσουμε και άλλα φάρμακα στη ρύθμιση ή όχι. Εμεί είμαστε ανοιχτοί τέλο πάντων για επαφέ με την Επιτροπή Περιβάλλοντο επ' αυτού, αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και θα σα τα πούμε. Thank you. E για το ECR. Commissioner, uh, in the last decade... Uh, την τελευταία δεκαετία, Επιτροπή, είμαστε μάρτυρες μια εκθετική αύξηση των σαρκοφάγων, των αγριόχειρων και άλλων αγρίων ζώων και άλλων ειδών που καταστρέφουν τη γεωργία. Μισό λεπτό λέει ο πρώτος γιατί προσπαθεί να, δει που κάθεστε. Ε, εκεί, εκεί, εκεί πίσω, αριστερά. Σηκώνει το χέρι ο κύριο Χιώκη. Αυτά λοιπόν ε, τα είδη έχουν και στη βιοπικιλότητα καταστροφικές επιπτώσεις, οπότε χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα δράσης ευρωπαϊκό. Οπότε να καλυφθεί και η βιοπικιλότητα με την ασφάλεια του κόσμου και τον οικόση των ζώων. Πέραν το ότι παίζεται η επιβίωση των μικρογεωργών και μικροαλλιέων. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε πει πολλές φορές θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία γιατί συνέχεια υπάρχουν ε, προβλήματα με αυτά τα είδη και ιδίως τους λύκους. Εσείς τι καθημερινές γραμμές θα δίνετε ως επίτροπος. Να έχουμε δηλαδή κάποιες εξαιρέσει στην περιβαλλοντική νομοθεσία, να δούμε τι θα γίνει με τις ποσοστώσεις ε, και πάρα πολλέ κοινότητε που εξαρτώνται από το ψάριμα έχουν πρόβλημα όσον αφορά αυτή την νομοθεσία. Έχουμε επίσης και τα νέα είδη, 25 εκατομμύρια υπολογίζονται, χώρα χαρακτηριστικά κλπ. Οπότε τι θα γίνει, ε, τι θα κάνετε επίσης και με τις περιοχές που έχουν ε, η μόλυνση. Ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω 100% τι είπατε. Στη δική μου χώρα, ξέρετε, υπάρχει η γεωργική δραστηριότητα και καταλαβαίνω ότι χάνουν τα κόστα ζώα τους οι γεωργοί. Οπότε το πρώτο είναι αυτό είναι να υπάρχει μια λύση δραστική, αλλά δεν είναι μαϊκή λύση. Αυτό που λέμε σημαίνει ασφαίρα. Αλλά είναι επικίνδυνη η κατάσταση με τους λύκους. Είναι θέμα συνύπαρξης. έκαθεν ήταν εκεί η λύκη. Προσπαθούμε απλώς αυτό να το σεβαστούμε, οπότε η συνύπαρξη επιτυγχάνεται με προστατευτικά μέσα. Προσπαθούμε να δούμε αν υπήρχε φράχτης, αν υπήρχε ικανή προστασία των οικόσιτων, ούτως ώστε να μην μπορεί να τα πιάσει ο λύκος. Άρα είναι θέμα συνειδητοποίησης, ε, ενημέρωσης του κόσμου, των γεωργών. Και έτσι θα το θέμα της ε, σύμπραξης παρόλα αυτά, ιδίως για τους βιότοπους και οι συναφείς που είναι ευέλικτες και έχουν περιθώριο τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των νομοθετημάτων. Οπότε, έτσι αυτή τη μέθοδο θέλουμε να ακολουθήσουμε κατανόηση, συνύπαρξη, προστασία των οικόστων για να λάβουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν και επιδοτήσεις από το πρόγραμμα LIFE για αυτές τις ενέργειες. Από την άλλη μεριά βέβαια για τα ζώα που χάθηκαν υπάρχει και μια ολική αποζημίωση επερώτηση. Για πετε μου τη γνώμη σας. Η οδηγία για τους βιότοπους μπας και δεν εφαρμόζεται αρμονικά και εναρμονισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το βλέπετε εσείς. Thank you, thank you for your question. First of all, I think, uh... Ο Επίτροπος, πρώτα-πρώτα. Η οδηγία έχει περάσει από το τεστ καταλληλότητας και είναι κατάλληλη η κρίθη. Υπάρχει ευελιξία που δίνει το περιθώριο στις χώρες να λύσουν τα θέματα εάν χρειάζεται. Και προστασία άλλων ειδών. Έχουμε 66 ήδη υποδικινές και δεν είναι μόνο οι αρκούδες και οι λύκοι, είναι και άλλα είδη και οπότε υπάρχει κάποια σύγκρουση ρυθμίσεων έχουν, έχουν, έχουν οι εθνικές αρχές την ευελιξία να το διαχειριστούν. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση για τον πρώτο γύρο των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την ΓΚΟΕ η κυρία Μπιόρκ. Εδώ είμαι κύριε υποψήφια Επιτροπέ. Έχετε πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, όπως είπατε. Όχι μόνο οι νέοι, αλλά και οι πολύ νέοι μας παρακολουθούν. Η κλιματική δικαιοσύνη, η βιοπικιλότητα είναι τα θέματα τα οποία θα κρίνουν το μέλλον μας και χρειάζονται συστημικές αλλαγές. Νομίζω ότι πολλοί από εμά ε, δεν ε, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει αυτές τις συστημικές αλλαγές. Όταν ακούω σχέδια δράσης, βλέπω πίνακες βαθμολογίες ε, και τον κίνδυνο να χαθούμε εδώ πέρα με στους λοιπόν. Το ερώτημα είναι το εξή. Δεν έχουμε αρκετά εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, ποια θα αναπτύξετε σε σχέση με άλλους ε, κλάδους με τους οποίου ανταγωνιζόμαστε, όπως η κοινή γεωργική πολιτική, η εμπορική πολιτική, η βιομηχανική πολιτική τη Ένωση. και να αλλάξουμε επίσης ε, τον τρόπο κατανάλωσης στην Ευρώπη. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα λοιπόν για τη βιοποικιλότητα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας και νομίζω ότι σωστά είπατε και δεν θα ξεχώριζα κάτι από αυτά. Όλα αυτά πάνε μαζί. Γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές και ενέργεια. Όλα είναι σημαντικά και προκαλούν απώλειες στη βιοποικιλότητα έχουμε έναν στρατηγικό στόχο. Είμαι σίγουρος ότι πιθανότατα θα χρηματοδοτηθεί καλύτερα. Αλλά τα λεφτά θα πάνε πεταμένα εάν δεν ε, περιληφθεί η στρατηγική της βιοπικιλότητας ε, και σε άλλους ε, τομείς. Και νομίζω ότι ε, αναφέρεται σαφώς ε, και στην επιτολή ανάθεσης ε, καθηκόντων του Αντιπρόεδρου Τίμερμανς ότι εγώ ως Επίτροπος βεβαίως πρέπει να έχω αποτελέσματα αλλά ο Αντιπρόεδρος θα φροντίσει, θα διασφαλίσει συντονίζοντας ότι θα ενσωματώνται και στους άλλους τομείς της πολιτικής. Έτσι θα επιτύχουμε αποτελέσματα και δεν θα έχουμε μόνο έτσι, πίνακες βαθμολογίες τους οποίους πρέπει να έχουμε για να μετράμε τα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει μέτρηση των αποτελεσμάτων, να υπάρχει λογοδοσία, αλλά όπως είπα να υπάρχει η πολιτική αυτή και στους άλλους ε, κλάδους που προκαλούν αυτή τη στιγμή την εξαφάνιση της βιοποικιλότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσετε κάποιες σοβαρές μάχες πριν φτάσουν αυτά τα θέματα στο γραφείο του Τίμερμαντς. Η στρατηγική από το χωράφι ως το πιάτο θα είναι ένα από τα εργαλεία σας. Πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να επηρεάσετε την κοινή γεωργική πολιτική για να έχει αποτελέσματα για την κλιματική δικαιοσύνη, για τον καταναλωτή και για την υγεία και την βιοποικιλότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα η στρατηγική αυτή από το χωράφιο στο πιάτο θα είναι εργαλείο για να σταματήσει η αποδάσωση και δεν μιλάω μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αξιολογήσουμε το αποτύπωμά μας και εκτός Ευρώπης και είναι σημαντικό που βλέπω εγώ την εντολή μου εδώ πέρα. Είναι η αλία για να γνωρίζουμε και να μπορούμε να εχνηλατήσουμε τα ψάρια από τα δίχτυα μέχρι την ε, κονσέρβα για να ξέρουμε τι μας ε, σερβίρουν εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε υψηλές προδιαγραφές. Και δεύτερον βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την αποδάσωση. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η αλυσίδα παραγωγής και αν επηρεάζει την αποδάσωση. Κύριε Οριστάντε Επίτροπε, ολοκληρώσατε τι αρχικέ σα παρατηρήσει λέγοντα ότι με πολύ μεγάλη χάρα θα συνεργαστείτε την επόμενη πενταετία με του βουλευτέ του Ευρωκοινοβουλίου. Ω Βρετανό, θα σα πω ότι μακάρι και εγώ να έχω την ίδια τύχη όπω εσεί. Έχουμε τώρα την ε, Επιτροπή Αλίας που θα πάρει τη σκητάλη. Ο πρώτος είναι ο κύριος Μιγιάν ε, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριο Ριστέντα Επίτροπε, εγώ ε, χαίρομαι για στην αρχή της παρέμβασής σας. Καταλάβατε ότι πρέπει να προσθεθεί η λέξη αλία στο χαρτοφυλάκιό σας. Και θέλω να το στηρίξετε το αίτημα αυτό και να το διαβιβάσετε και στην Πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Και τώρα, αν με επιτρέπει ο Πρόεδρος, να αναφερθώ ακριβώς και εγώ στο Brexit. Δεν πιστεύουμε πολύ η οικονομική εταιρική σχέση που θα θεσπιστεί στο μέλλον μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου θα συνοδεύεται και από μια συμφωνία που θα ε, διατηρεί την αμοιβαιότητα στην πρόσβαση στα ύδατα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σα. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Πρέπει να υπάρξει διαγενειακή ανακύκλωση στην Αλία. Είναι κάτι που το θέλουμε. Για να προσελκύσουμε τους νέους πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και όχι να υπάρχει υπεραλίευση. Δεν μιλώ γι' αυτό. Θέλουμε καλύτερη αλία. Και νομίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις. Ποια είναι η άποψή σας ε, για την αλλαγή σκητάλης μεταξύ των γενναιών λοιπόν, που είναι σημαντικό θέμα. Και έρχομαι στην ε, βιοτεχνική, τη μικρή κλίμακα παράκτη αλία, 75% ε, δύσκολα προσαρμόζεται στις αλλαγές, στις βίες αλλαγές αυτός ο κλάδος και θα πρέπει να το λάβετε υπόψη στις νομοθετικές αλλαγές που ενδεχομένως προωθήσετε, να γίνουν μελέτες αντικτύπου και να εφαρμόζονται βαθμιδών αυτές οι τροποποιήσεις ε, στην παρακτιαλία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το Brexit, χτες ε, κατατέθηκε μια πρόταση, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς αν και πότε και πώς θα συμβεί το Brexit. Ναι, κάποιο σχόλιο εκτός μικροφώνου, ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να πω ότι είμαι ευγνώμων στον κύριο Μπαρνί γιατί προσφέρθηκε να με συναντήσει δύο εβδομάδες, επόμενες δύο εβδομάδες για να συζητήσουμε. Και φυσικά θα συζητήσουμε και με τη Μεγάλη Βρετανία για το οποιοδήποτε σενάριο. Σίγουρα θα υπάρξουν ε, διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις πάνω σε ένα Brexit με συμφωνία, γιατί αυτό θα είναι πιο εύκολο, θα υπάρχει μεταβατική περίοδος, ε, ενώ αν δεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία θα να συζητήσουμε εν συνεχεία. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι, να είστε βέβαιοι ω προ αυτό. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων και την ε, ανακύκλωση των γενεών. Στο Στρασβούργο τα έχουμε πει. Έχω επίσης ε, μιλήσει με άλλους Ισπανούς βουλευτές και Ιταλούς βουλευτές που έχουν θέσει το ίδιο θέμα. Και πραγματικά με έχει απασχολήσει το θέμα. Παραδείγματο χάρη, αν βελτιωθούν ε, οι συνθήκε πάνω στα σκάφη, θα προσελκυστούν περισσότεροι νέοι. Τι να σα πω, ειλικρινά δεν είμαι και τόσο σίγουρο. Γιατί και εγώ νέο είμαι αν έπρεπε να διαλέξω ποιο θα ήταν το βασικό στοιχείο που θα επηρέαζε την επιλογή μου, εγώ νομίζω η ασφάλεια για το μέλλον μου. Αυτό θα ε, ήταν ε, ο γνώμονας. Άρα θέλουμε αυτό να εξασφαλίσουμε και πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ κοινωνικών, οικονομικών ε, παραμέτρων και βιωσιμότητας για να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον στον τομέα αυτό και με τη χρηματοδότηση από το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και από άλλες πηγές μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να βελτιώσουμε τις αλείς και τους αλείς διακόπτεται ο Επιτρόπος. Uh, Επερώτηση από τον κύριο Μιγιάν Σα ευχαριστώ που δεσμεύεστε για την αλλαγή σκητάλη μεταξύ των γενών. Είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για το μέλλον. Επίση, οι καλέ συνθήκε διαβίωση και συνθήκε εργασία πάνω στα σκάφη είναι κάτι σημαντικό για να είναι πιο ελκυστικά τα ναυτικά επαγγελμάτα. Τώρα, για το Brexit, δεν έλεγα αν θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει και τι μεταβατική περίοδο θα έχουμε. Αλλά λέω, ποια θα είναι η μελλοντική σχέση μετά το Brexit. Θέλω να είναι φιλόδοξη αυτή η εταιρική σχέση. Θα είναι μόνο οικονομική εταιρική σχέση. Δεν θα πρέπει πρέπει να θυσιάσουμε την αλία σε μια μεγάλη οικονομική εταιρική σχέση που θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να περιληφθεί μια διμερής συμφωνία για να υπάρχει πρόσβαση αμοιβαία σε πόρου και ύδατα. Πάνω σε αυτό σα ρωτούσα. Ποια θα είναι η μελλοντική σχέση σε περίπτωση Brexit. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Και συμφωνώ σε ό,τι αφορά τους νέους ότι μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και ελπίζω να έχουμε διάλογο θα καλέσουμε τους ενδιαφερομένους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είναι ένα ευγενές επάγγελμα αυτό του Αλιέα. Τώρα για το Brexit, φυσικά και θα υπάρξει μετά το Brexit μια σχέση ε, και φυσικά δεν πρέπει να αποκλείουμε την Αλία, θα υπάρξει συμφωνία. Ε, ο κύριος Μπαρνιέ, σα το λέω ξεκάθαρα, θεωρεί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα γιατί διατέλεσε στη Γαλλία Υπουργός Αλίας, γνωρίζει τα προβλήματα Άρα είναι καλυμμένο αυτό το θέμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος γι' αυτό. Ενάμιση λεπτό κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε υποψήφιε. Ο ληφτικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας, τη γαστρονομία, την πολιτιστική ταυτότητα και την ασφάλεια των τροφίμων για πολλές παράκτες περιοχές αντιπροσωπεύει μέχρι και το ίμιση των θέσεων εργασίας. Των θέσεων εργασίας λοιπόν στις μικρές περιοχές αυτές τις παράκτες και η χώρα μου η Ισπανία δίνει μεγάλη σημασία και δυστυχώς θα επανέλθω και εγώ στο ότι δεν αναφέρεται καν η λέξη αλία σε κανένα χαρτοφυλάκιο, σε, στον τίτλο κανενός χαρτοφυλακίου. Αυτό εμάς μας ανησυχεί. Τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για και την Αλία. Εμείς ζητούμε να μην υπάρξει περικοπή καμία της χρηματοδότησής του. Ελπίζω να το προωθήσετε, γιατί πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και έχουμε και την κοινωνικο-οικονομική διάσταση, που είναι επίσης ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της αλληλευτικής πολιτικής και ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος και η παράκτη αλληλεία. Και ένα σημαντικό θέμα που πρέπει εσείς να το έχετε υπόψη σα είναι ακριβώ οι νέοι και πώ την κοινωνικο-οικονομική διάσταση τη αλληλευτική πολιτική θα την εξασφαλίσετε και τα πολυετή προγράμματα. Πράγματι, μεταξύ των διαφόρων λεκανών υπάρχει μεγάλη ε, ποικιλία, πολυμορφία. Τι θα κάνετε λοιπόν, ιδίω για την Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Thank Thank you for your question. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά τις παράκτιες ε, περιοχές και κοινότητες, φυσικά και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Είμαι ακόμα υπουργό ε, Οικονομής και Καινοτομία ε, και όταν ε, ανέλαβα καθήκοντα για μια διετία, τι έκανα κάθε Παρασκευή, πήγαινα σε μια διαφορετική περιοχή στη Λιθουανία. 60 συνολικά. Μέχρι τώρα έχω επισκεφθεί τις 52. Και όχι γιατί κάποιος με κάλεσε, αλλά γιατί με νοιάζει, ενδιαφέρομαι. Έχω επισκεφθεί επαγγελματικά, βιομηχανικά κέντρα και τοπικά καταστήματα, μικρά. Γιατί θέλω να δω ε, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι, τους οποίους ψηφίζουμε, αλλά πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται. Και ήθελα να το κάνω και με τους ψαράδες και είπα ότι θα έχουμε διάλογο. Η κοινή ελευτική πολιτική ακριβώς αυτό θέλει να πετύχει. Ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας και των κοινωνικονομικών πτυχών. Και το Ταμείο για τη θάλασσα και την Αλία, φυσικά είναι ένα εργαλείο, είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Σε ό,τι αφορά τα πολιετή προγράμματα, Φυσικά και κάθε, λεκάνη, ε, κάθε θαλάσσια λεκάνη είναι ξεχωριστή και πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Θα πρέπει να λάβουν πώ τα γνωμοδοτικά συμβούλια επίση, ε, για να δούμε ποιε είναι οι θέσει των κρατών μελών και έπειτα να καταλήξουμε ε, σε σχέδια ισορροπημένα, εξασφαλίζοντα τη βιωσιμότητα αυτό είναι το μακροπρόθεσμο στίχημα και έτσι θα προσελκύσουμε τους νέους στον κλάδο. Συμφωνώ, η ασφάλεια είναι κάτι σημαντικό. Οι συνθήκες εργασίας είναι σημαντικές και αυτές. Συμφωνώ. Αλλά οι νέοι πρέπει να βλέπουν ότι τους δίνει μέλλον για αυτούς και για την οικογένειά τους αυτό, αυτή η απασχόληση, ότι μπορεί να έχουν κέρδος και ότι μπορεί να έχουν μια σταδιοδρομία, μπορεί να διευρύνουν ε, τη δραστηριότητά τους και το στόλο. Sí, me gusta que αναγνωρίζετε την ε, σημασία και του κοινωνικού, οικονομικού και του περιβαλλοντικού πυλώνα, έτσι. Είναι καλό γιατί δεν το αναγνωρίζουν όλοι. Αλλά ε, μια διευκρίνηση ε, σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο. Θα μας υποστηρίξετε για να μην περικοπούν τα κονδύλια της αλίας. Είναι ένα μικρό τάμιο αυτό τη και χρειάζεται όλου του πόρου που μπορεί να έχει. Και τέλο, τι θα κάνετε για το ρόλο τη γυναίκα ε, στον αλληλευτικό τομέα που τι περισσότερε φορέ ούτε καν αναγνωρισμένο είναι, πόσο μάλλον ρυθμισμένο. Και ο προκάτοχό σα ε, δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα αυτό. Ε. Σα παρακαλώ λοιπόν να κάνετε εσεί ό,τι μπορείτε. Uh... Σα ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το MFF, ε, την πρόταση την έχετε επιτάπητος ε, για το Ταμείο αυτό και ελπίζω να είμαστε φιλόδοξοι. Ε, υπάρχει σίγουρα η διάσταση της βιωσιμότητας ε, και η περιβαλλοντική κοινωνικο-οικονομική διάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις γυναίκες και την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Δυστυχώς, είδα την τελευταία έκθεση του ΒΒΕΦ και πραγματικά πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μην εστιάζουμε μόνο ε, στο ψάρεμα αυτό καθεαυτό, γιατί φυσικά εκεί τη δουλειά την κάνουν πιο πολλοί άνδρες, αλλά είναι ένα ε, μόνο από τα επαγγελματά από πίσω, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Και ποιος έχει να κάνει με τις ε, επαφές, με τα διάφορα κρατικές αρχές, με τα οργάνωση. Όλα αυτά τα κάνουν πολλές γυναίκες, πολύ μεγάλο βαθμό γυναίκες. Άρα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή, να υπάρχει σε εκπροσώπηση. Και είπα και εγώ ότι πρέπει να εμβαθύνουμε, πρέπει να συζητήσουμε με τον τομέα. Και όχι μόνο του μεγάλους, αλλά και τους μικρούς. Ευχαριστώ, κύριο Κάρλες Κίντ, 1,5 λεπτό. Ε, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, η τελευταία μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής το 2013 μας έδωσε διάφορα μέσα άσκηση αυτής της πολιτικής, του ε, μέσο για τις εκφορτώσεις και άλλα τεχνικά μέτρα, επί όσον αφορά τον ε, γόνο και την αλία του ε, και σε σχέση με κάποια βιώσιμη διαχείριση στον αφορά περιβάλλον, αλλά ε, οι στόχοι ήταν πολύ πιο φιλόδοξοι. Να με την Βαλτική που την ξέρετε. Είχαμε ένα πρόγραμμα εδώ και τρία χρόνια, αλλά είδαμε ότι τα αποθέματα του μπακαλιάρου έχουν πέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι βέβαια θέμα η μόλυνση αλλά και η αλλαγή του κλίματος. Έχετε ένα χαρτοφυλάκιο πολύ πλούσιο και πώς το βλέπετε τα πράγματα, τι θα γίνει για τα οικοσυστήματα, τι θα γίνει για τους ελληνικούς πόρους, τι μπορεί να γίνει για μια βιώσιμη γεωργία με το 2030. Θα μετέλθετε όλα τα θέματα που έχετε για να καλύψετε όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν ε, τους αλληλευτικούς πόρους. Ο Επίτροπος, σας ευχαριστώ. Ναι. Η βιομάζα μειώνεται από, τη, από την αλία, το ίδιο και η ελευθερική πόρη και έχουμε βέβαια την στρατηγική όχι μόνο για την ξηρά αλλά και για την θάλασσα της θάλασσας και τους ωκεανούς που θέλουμε να διέπονται από υγεία. Εκεί απορροφάται πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακος, οπότε βοηθούμεθα και στο ενεργειακό και στην απασχόληση. Τέτοια ε, κοινή πολιτική θέλουμε, όπως έγινε και η μεταρρύνηση του 13 Και οπότε Μέχρι το 22 θα κάνουμε μια άλλη αναθεώρηση, θα διορθώσουμε τα κακοσκήμενα, αλλά να είμαστε ρεαλιστές, η κοινή πολιτική δεν είναι μια γενική σφαιρική νομοθεσία που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Από τώρα, με στρατηγική βιοπικιλότητα θα πρέπει να τα διορθώσουμε τα κακοσκήμενα και το Green New Deal θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλές μεταβλητές. και τις νέες πρόκλησεις, άρα να προχωρήσουμε με προσοχή με τον ορίζοντα του 2022 και θέλουμε την βοήθεια του Κοινοβουλίου γιατί το θέμα είναι πολύ τεχνικό και δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, υπάρχουν και ζητήματα κοινωνικά. Άρα Γι' αυτό και υπολογίζω στη βοήθειά σας, πραγματικά. Έπερα του κ. Καρλίσκιν... Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα που το πάτε και μπράβο το ότι θέλετε να πηγαίνετε επί τόπου να συναντάτε τον κόσμο τους ενδιαφερόμενους. Μπράβο. Τώρα, εγώ προτείνω όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν και που θα κάνετε και εμείς θα τις ε, υπερψηφίσουμε θα πρέπει όλα αυτά να τα θεσπίσουμε από κοινού, να το κάνετε με εμά και όχι μόνο με τους υπαλλήλους σας. Εμείς επίσης εκπροσωπούμε τον κόσμο. Πρότασή μου είναι να μην έρχεστε μια φορά το χρόνο εδώ. Να έρχεστε να τα λέμε επισήμως και ανεπισήμως εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρλσκιν για την πρόσκλησή σας. βεβαίως και όπως είπαμε για το Στρασβούργο και για την Βρετάνη θα κάνουμε μαζί την επίσκεψη και υπολογίζω στην συμπαράσταση σας. Η κυρία Σάλιβαν και τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον υποψήφιο Επιτροπό. Το ερώτημά μου αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ε, και Θαλάσσης. Η συζήτηση για το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα το γεγονός ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπεραλλιεύει όπως μας δείχνει η τελευταία αξιολόγηση της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής 49% των αλλιευμάτων στον Βόρειο-Ανατολικό Ατλαντικό υπεραλλιεύονται. Η βελτίωση είναι λίγη και γίνεται πάρα πολύ αργά. Βλέπουμε ειδικά ε, στην ε, Μεσόγειο πως ένα 87% των ηχθείων αποθεμάτων των ειδών υπεραλλιεύεται. Και με το πι μπορεί να έχουμε αύξηση της δυναμικότητας του τομέα σε αντίθεση με τους δηλωμένους στόχους της ε, πολιτικής αλίας της Ένωσης οι επιδοτήσεις οδηγούν στην υπεραλία και δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα. Υπάρχουν εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εξηγούν το πρόβλημα με όρους δραματικούς. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι το εξής. Τι θα κάνετε έτσι ώστε η θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους που έχουμε συμφωνήσει για την βιώσιμη ανάπτυξη και τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ για να απαγορευθούν οι καταστρεπτικές επιδοτήσεις που αυξάνουν τη δυναμικότητα του στόλου. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Συμφωνώ. Το ΠΔΠ πρέπει να υποστηρίζει τους στόχους μας. Ε, εφαρμογή της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, ε, δεσμεύσεις για την εφαρμογή των, ε, του στόχου 14, του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, βεβαίω ο φάκελος αυτός δεν είναι απεριόριστος και πρόκειται για χρήματα του φορολογούμενου. Ως πρώην Υπουργός ε, Οικονομικών και Γενοτομία στην Λιθουανία, είχα ένα τεράστιο ποσό ε, κοινοτικής χρηματοδότησης. Ο βασική μου αρχή ήταν να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη με την ιδιωτική χρηματοδότηση. Αν βλέπουμε ότι κάποιοι τομεί μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ιδιωτική χρηματοδότηση, δεν θα ξοδέψουμε δημόσιο χρήμα. Γιατί δεν υπάρχει αρκετό. Βεβαίω, δεύτερον, ελπίζω να διατηρηθεί η φιλοδοξία και οπωσδήποτε θα είμαι στην διάθεσή σας για διάλογο στην Επιτροπή να διατηρηθεί αυτή η φιλοδοξία μαζί με τα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνομαι τις ε, ανησυχίες τους και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να δούμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Η... των μικρών αλλιέων. Αλλά όπως σας είπα δεν μπορεί να είναι σε αντίση με τους ε, στόχους μας ε, για την αλληλεία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αυτό ήθελα να πω είπατε ότι δεν θα επιτρέψετε η πολιτική της Ένωσης ε, να είναι αντίθετη με τα επιστημονικά δεδομένα και αντιλαμβάνομαι ότι είστε διατεθειμένος και αυτή είναι η ερώτησή μου θα είστε διατεθειμένος να αποσύρετε μία πρόταση χρηματοδότησης εάν αντιβαίνει την ορθή πολιτική βιωσιμότητας. Σας ευχαριστώ. Ας μην βιαζόμαστε για περικοπές και κόκκινες γραμμές γιατί κάποιος ε, θα φέρει μετά μια αντίρρηση και θα πρέπει να απαντήσουμε αναλόγως. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο για τα ζητήματα. Συμφωνώ ότι τα χρήματα του φορολογούμενου πρέπει να εξοδεύονται για να επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Σημαντικό επίσης είναι ότι ζούμε σε ευαίσθητη περίοδο. Μπορεί να συμβεί το Brexit και βεβαίως θα έχει ε, ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και θα ξεκινήσει το 2021. Οπότε δεν είναι ανοιχτή και υπεραιτέρω καθυστέρηση του. Οπότε Πρέπει να εκθέσουμε τα επιχείρηματά μας και να βρούμε την καλύτερη λύση, να επιτύχουμε μια ισορροπία. Κυρία Κόντε, για την ομάδα ID 1,5 λεπτό. Ε, για να σας βλέπει και ο Επίτροπος. Κύριε Συγκεβίτσιους, από το 1977 μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει 11 επίτροποι στην δική σας ε, θέση και πάντα βεβαίως η αλληλεία ανήκε στο χαρτοφυλάκιο των προκάτοχων σας. Σήμερα έχουμε ένα γενικόλογο περιβάλλον και ωκεανή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυρία Φόντερ Λάιν δεν αποδίδει αρκετή σημασία σε αυτόν τον πολύ σημαντικό οικονομικό τομέα. Είναι προφανές πως η Κομισιόν δεν έχει καταλάβει την θεμελιώδη σημασία του κλάδου αυτού. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από εσάς, όταν έχετε καταργήσει και την λέξη αλληλεία, θα καταργηθεί η στήριξη του κλάδου. Θα πρέπει να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των ε, ψαράδων. Θα πρέπει να αποκατασταθεί λοιπόν η προσοχή, η αξία της ε, αλίας. Μιλάμε πράγματι για τους ε, πόρους, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαστούμε τον ένα νόμο με τον ε, άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω το εξή: Σκοπεύετε εσείς να αυξήσετε, να μειώσετε ή να διατηρήσετε σταθερούς τους πόρους για την ε, αλληλεία. Θα επιμείνετε στην ονομασία του χαρτοφυλακίου σας ε, ή θα θελήσετε να αλλάξει και να ονομαστεί για, την, για τους ωκεανούς και την αλληλεία. Ευχαριστώ. Thank you for your Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα για την ονομασία του χαρτοφυλακίου. Ας πάμε παραπέρα από το όνομα, ας δούμε την ουσία. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπορείτε ε, να με αξιολογήσετε σήμερα αν θα βοηθήσω τις ε, κοινότητες ή όχι. Ε, δεν ε, θα τα κάνει αυτά το όνομα του χαρτοφυλακίου. Πρέπει να δούμε σήμερα το τι απαιτείται για τους ψαράδες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Και πολύ σωστά παρατηρήσετε ότι υπάρχει μια πρόταση για τη χρηματοδότηση ε, η οποία ε, δεν θα αλλάξει, υπάρχει ήδη, συζητείτε. Αλλά είναι επίσης ε, σημαντικό να βοηθήσουμε και τους ψαράδες να αντιμετωπίσουν και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να αντιληφθούν ότι η μείωση της βιομάζας δεν είναι μόνο θέμα αλίας, Είναι πολύ ευρύτερο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί. Να μην διαχωρίζουμε το περιβάλλον από την αλία. Αυτά πάνε μαζί. Το υγιές περιβάλλον έχει και υγιή ψάρια, μεγαλύτερα ψάρια. Μεγαλύτερα ψάρια σημαίνουν περισσότερα κέρδη για τους ψαράδες και τις παράκτης κοινότητες. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και να προσπαθούμε να τον ε, επιτύχουμε μαζί. Μην ξεχνάτε όμως, ε, παρά το ότι δεν υπάρχει στο όνομα του χαρτοφυλακίου σας, ε, το υπεύθυνο μέλλον της αλληλείας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να τονίσω την δύσκολη κατάσταση της αλληλείας στην Μεσόγειο. και θα πρέπει ακριβώς ε, να δούμε πώς οι παράκτητες κοινότητες αντιμετωπίζουν την μείωση των ε, αποθεμάτων και άλλες ε, προκλήσεις. Γι' αυτό σας ερωτώ, τι στρατηγική θα αναμένουμε για την Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να έχουμε ίσους όρους ε, ανταγωνισμού και να σταματήσει η ε, παράνομη αλία γιατί οι μικροί ψαράδες έχουν, αυτοί έχουν τα, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με την παράνομη αλία και η παράνομη αλία δεν είναι μόνο θέμα του ότι πιάνονται ψάρια είναι και ε, προβλήματα οικονομικά, δεν πληρώνονται φόροι, δεν υπάρχουν οι όροι ασφαλείας ε, κτλ. Οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Τώρα για την εμπιστοσύνη που είπατε. Πριν από την ακρόαση, ε, επισκέφθηκα εδώ τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και το αστείο με την ε, συνθήκη της ε, Ρώμης το 1957 ε, υπογράφηκε στην πρώτη σελίδα και στις τελευταίες σελίδες. Λοιπόν, έχει οικοδομηθεί η κοινότητα στην εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. θα ήθελα να απαντήσετε και σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Κόντε για την Μεσόγειο, η οποία είναι και μία από τις πιο υπεραλλιευμένες θάλασσες στον κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Έχει υπάρξει μια πρόοδος όσον αφορά τα πολιετή σχέδια στην ε, Μεσόγειο. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία αυτή να αξιολογήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα από θέματα γιατί δεν αξιολογούνται σωστά. Και αν έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, τότε θα έχουμε μια σωστή προσέγγιση για την ε, βιωσιμότητα για τους ψαράδες. Επίσης, σημαντικές είναι οι διμερείς συμφωνίες, όπως ε, οι συμφωνίες με τις άλλες χώρες της ε, Μεσογείου. να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να φροντίσουμε ότι δεν θα σεβόμαστε μόνο εμείς ε, τους ε, νόμους, αλλά και οι εταίροι μας. Σας ευχαριστώ κυρία Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, η περιφερειοποίηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο είναι προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη και με την κοινή ελληνική πολιτική. Προβλέπεται περιφερειακή συνεργασία για την προστασία της θάλασσας, για τα πολιετή προγράμματα και για τα προγράμματα που αφορούν τις απορρίψεις. Εσείς θα το εξασφαλίσετε αυτό θα είναι στους νομοθετικούς σας στόχους, ιδίω όσον αφορά ακριβώς την προετοιμασία νομοθεσιών ή μάλλον προγραμμάτων για την πελαγική αλληλεία. Περιφερειακή συνεργασία. Να μην έχουμε πια κενά στην νομοθεσία, στα προγράμματα, γιατί για τα μικρά πελαγικά ψάρια, στην Αδριατική, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα πολύ μεγάλο να λαμβανθεί υπόψη η ιδιορυθμία της Αδριατικής αλλά και της Μεσογείου. Thank you. Indeed, I think, as you said, every sea basin is unique and it... Ακριβώς. Κάθε θάλασσα έχει τα χαρακτηριστικά και χρειάζεται αυτό να σταθμίζεται, οπότε βέβαια το κλειδί είναι βέβαια να πετυχαίνουμε την βιωσιμότητα. Στη Λιθουανία εξελέγει ω βουλευτή. Άρα πιστεύω στο διάλογο και τα πολιετή προγράμματα ακριβώς αφορούν τον διάλογο να εμπλέκονται οι αλλοίς και να υπάρχει διάλογος και με τρίτες χώρες για εξέβρεση των εφικτών λύσεων. Σε αυτή τη ρότα πρέπει να συνεχίσουμε. Τα πολιτικά προγράμματα έδειξαν ότι υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την υπεραλίευση των πόρων και με τις σχετικές συμφωνίες θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Άρα και μεταξύ κρατών μέλων και με τρίτες χώρες να έχουμε συμφωνίες. Ερώτηση. Θα ήθελα ακόμη να μου πείτε πώς θα εγγυηθείτε τα σχετικά αποτελέσματα αυτά τα, τις συμβουλευτικές επιτροπές, αυτά τα γνωμοδοτικά συμβούλια θα τα λάβετε υπόψη. Θα εξασφαλίσετε την περιφερειοποίηση και την επαρκή αντιπροσώπευση όλων των εμπλεκομένων. Ο Επίτροπος. Ε, βέβαια. Για τα γνωμοδοτικά συμβουλιά τόσα χρόνια. Ήταν αξιόπιστοι συνεργάτες μας, εταίροι μας. Για τον τόνο, για τη μετακίνηση, μετανάστευση του τόνου. Ε, βέβαια. Και η συνεννόηση θα συνεχιστεί. Ακριβώ αυτή είναι η δουλειά των συμβουλίων αυτών και εκπροσωπούνται και οι μεγαλοαλείς και οι μικροαλείς. Κύριε Σενκεβίτσιος, εδώ, εδώ, εδώ κάθομαι. Πριν από μερικέ μέρε είχαμε την δημοσιοποίηση μια έκθεση πολύ ενισχυτή για του ωκεανού. μεγάλη η μόλυνση, ασφυξία. Από το 50, 77 δις τόνων οξυγόνου εξαφανίστηκαν. Τι θα κάνετε για την εντατική χθιοκαλλιέργεια και την υπόλοιπη μόλυνση. Τα σόναρ, οι θαλάσσιες μεταφορές, και ιδίως τα θαλάσσια κήτη κινδυνεύουν. Δεν πρέπει τα βαπόρια να ταξιδεύουν πιο αργά και να υπάρχει προστασία κάποιων ζωνών. Τι γίνεται με τον τουρισμό στους πόλους. Αυτό γίνεται και από τα χρησιμοποιημένα βρώμικα ύδατα, από τα χωροκατακτητικά, ήδη από τα φύκια. Δεν πρέπει να εκεί να μειωθεί, να περιοριστεί ο τουρισμός να υπάρχουν επίσης λιγότερο βλαπτικά κάψιμα. Να γίνει κάτι σε σχέση και με τα όσα έχει εξαγγείλει ο ΙΕ για την προστασία των θαλασσών. Να προσχωρήσουμε σε αυτή την ε, συμφωνία του ΙΕ. Okay. Thank you very much for your question. ευχαριστώ. You're absolutely right. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντική η ωκεανία και είναι σημαντικό να του προστατεύσουμε. Σημασία για τι παράκτε κοινότητε, για τους αλληλείς και ξέρουμε το τα βασικά θέματα, τη βασική αιτία του κακού είναι η υπεραλίευση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν προστατεύονται αρκετά. Έχουμε όλα αυτά τα σκουπίδια της θάλασσας και θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο διεθνές. Και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο το σέβονται όλοι και όχι μόνο εμείς. θα εκεί για την βιοπηγηλότητα του 2030 και είναι σημαντικό εκεί να καλυφθούν και οι ωκεανοί. Δεύτερον, η κυκλική οικονομία, όταν μιλάμε για τα απορρίμματα στη θάλασσα, όταν μιλούμε για τα φορτία αποβλήτων, ε βέβαια, είναι ευκαιρία για την οικονομία μας. Και στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, οι πόροι που αναλώνουμε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη λύση των προβλημάτων και να κάνουμε και πολλά άλλα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδυαστούν και οι προσπάθειες στο μέτωπο της γεωργίας όπως την ε, Βαλτική. Έχουν προβλήματα από απόβλητα μη βιώσιμα από την γεωργία. Επομένως όλες οι αιτίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά τα έχω στο χαρτοφυλάκιο και θεωρώ ότι είναι βασικό μου καθήκον. Για μένα αυτό ήταν καλό ότι όλα αυτά τα βάλαμε στο ίδιο χαρτοφυλάκιο αλληλεία, ωκεανούς, περιβάλλον, όλου αυτού τους τομείς που είναι αλληλένδετοι. Επερώτηση. Ευχαριστώ για την απάντηση. Συμφωνώ 100%. Δεν μπορεί μόνο να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι και για την Μεσόγειο που αγαπώ και πολλοί από εμά την αγαπούμε, πάρα πολύ μεγάλη εκεί πέρα η μόλυνση. Έχουμε τέσσερις φορές περισσότερη μόλυνση από πλαστικά από τον ειρηνικό. Ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι μέσω τη Ένωση για την Μεσόγειο για να, κάνουμε, να λάβουμε συγκεκριμένη δράση όσον αφορά τη μόλυνση στη Μεσόγειο. Thank you very much. Uh, Α, μάλιστα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Επίτροπος, για την Μεσόγειο. Ε, βέβαια πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και όχι μόνο στο να την καθαρίσουμε με ό,τι μέσα έχουμε με τις καλύτερες πρακτικές αλλά να το κάνει αυτό και η ελληνική πολιτική να καταπολεμήσουμε την παρανομία αλληλεία και επομένως έτσι θα πιάσουν τόπο οι πόροι μας να βοηθήσουμε και τους εταίρους μας να χτυπήσουμε την ρίζα του προβλήματος, να δώσουμε συμβουλές με τις πρακτικές μας και να συνεργαστούμε. Ε, βέβαια είναι σε θέση να καταστεί πρωτοπόρα η Ένωση σε αυτό το μέτωπο. Λοιπόν, περνάμε στον δεύτερο γύρο της ακρόασης, ε, κύριε υποψηφίου επίτροπε θα ακούσουμε τις υπόλοιπες 11 ε, ερωτήσεις σύμφωνα με τον κανόνα Ντεόντ και θα ε, είναι αλλάξει οι επιτροπές όχι από τη μία περιβάλλοντος και από την άλλη αλληλείας. Οπότε ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Κύριος Μαζίλης. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα να ε, επανέλθω στην απάντησή σας για τους λύκους. Οι αριθμοί τους αυξάνονται 13 έως 14.000 ε, ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία και η κτηνοτροφία υποφέρει. Και το ίδιο ισχύει με διάφορα πουλιά, όπως η Κορμοράνη. Και οι αλληλείς λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε επίπεδο που αποτελούν πλέον απειλή για την αλληλεία. Αυτό ισχύει και για την Βαλτική και τη Λιθουανία. Συμφωνείτε ότι απαιτείται περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να ρυθμίζουν τους πληθυσμούς κάποιων προστατευόμενων ειδών. Αν μου επιτρέπετε, μια που είμαστε συμπατριώτες, ε, θα μιλήσω την ε, γλώσσα μας. Σας ε, ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την ερώτησή σας. Είναι πολύ επίκαιρη η ερώτηση, αναφέρθηκε ήδη. Και η οδηγία την οποία αναφέρατε ε, προβλέπει ε, μια ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες ε, χάνουν το ψωμί τους, αλλά δεν λύνεται με βία μέσα με σφαίρες αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε αν έχουμε λάβει αρκετά μέτρα για να προστατευτούμε από τους λύκους. Ο φράχτης που είπα και πριν. Ε, μέτρα τα οποία μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ζημία που προκαλούν ε, στα ζώα και εκεί πέρα προβλέπεται αποζημίωση. Τώρα για τους κορμοράνους που αναφέρατε. Αποτελέσματα τα βλέπουμε ξεκάθαρα και στην ε, Λιθουανία, στην ε, θάλασσα εκεί. Και βεβαίως θα ήμουν υπέρ ε, μιας ρύθμισης για να ληφθούν ανάλογα μέτρα στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Για τις ε, παράκτιες ε, περιοχές, ε, εγώ είδα κορμοράνους στο Κάουνας που απέχει 200 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Δεν υπήρχαν κορμοράνοι στο Κάουνας. Σύμφωνα με την οδηγία η εσκεμμένη θανάτωση τέτοιων ε, ειδών ε, απαγορεύεται και τιμωρείται. Απ' την άλλη, πλήττονται εδώ πέρα τα συμφέροντα των ψαράδων ε, σε μεγάλο βαθμό. Και οι απειλές, και απειλείται και η βιοπικιλότητα. Θα θέλαμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, απάντηση. Θα ήθελα ε, να πω. Εδώ επανερχόμαστε στην ε, οδηγία. Ίσως η οδηγία πρέπει να επανεξεταστεί. Η Επιτροπή ήταν ε, εναντίον, όμως και εγώ το ίδιο θεωρώ, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε εάν ε, τα κράτη-μέλη εκμεταλλεύονται αρκετά την ε, ευελιξία που υπάρχει. Και βεβαίως ε, αν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή και πρόβλημα για τους ψαράδες όπως αναφέρεται, μπορεί να υπάρξει μια ευελιξία. για τους ε, σοσιαλδημοκράτες ε, η κυρία Μπουρκχατ. Σήμερα μιλήσατε για την ε, βιοπικιλότητα και σωστά μιλήσατε για μαζική εξαφάνιση των ειδών. Ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών απειλείται με εξαφάνιση. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγική της για την βιοπικιλότητα δεν θα επιτύχει τους στόχους της μέχρι το 2050. Με βάση αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα αναπτύξετε φιλόδοξους και δεσμευτικούς ε, στόχους ε, για την ε, βιοπικιλότητα μέχρι το 2030 και αν έπιους κατόπιν θα φροντίσετε να υπάρξει και το απαραίτητο προσωπικό και τέλος ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για τις ε, μέλισσες. Παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην επικονίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα, είχαμε στόχους για το 2010, για το 2020 Οπωσδήποτε θα έχουμε στόχους και θα είναι φιλόδοξοι γιατί δεν γίνεται αλλιώ και για το 2030. Δυστυχώς οι στόχοι δεν αρκούν. Πρέπει να ε, υπάρχει μέτρηση και παρακολούθηση. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τις βασικές αιτίες είναι η αλλαγή της χρήσης γης και θάλασσας, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, και τα χωροκατακτητικά είδη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αιτίες και όπως ανέφερα στην αρχή και σωστά σημειώσατε, αυτό σημαίνει ε, πράγματι χρηματοδότηση. Επανεισαγωγή ειδών ε, Natura 2000, αλλά δεν αρκεί. Και ελπίζω σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς να επιτύχουμε αυτόν τον ε, φιλόδοξο στόχο της ε, βιοπικιλότητας ε, του 2030. Οι στόχοι αυτοί περιέχονται και σε άλλα νομοθετήματα όπως της γεωργίας, βιομηχανίας, μεταφορών. Πρέπει να χρησιμοποιούμε λοιπόν τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Η αξιολόγηση αντικτύπου πρέπει να γίνεται πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, καμιά φορά έχουν εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη, όπως βλέπουμε, προσπαθούν να την ε, παρακάμψουν και αυτό δεν είναι ορθή πρακτική, ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές Natura 2000, όπου έχουμε πολλά προστατευόμενα είδη. Σας ευχαριστώ για την συγκεκριμένη απάντηση. Μιλήσατε για μετρήσιμους ε, στόχους, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος ε, με τι στόχους θα πάτε στη διαπραγμάτευση. Και το δεύτερο, είπατε πολύ σωστά ότι οι στόχοι από μόνοι τους δεν αρκούν. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για την τήρηση των όρων αυτών, να αυξηθεί η προστασία στις περιοχές ε, Natura και να υπάρξει αποκατάσταση των υποβαθμισμένων ε, οικοσυστημάτων. Σας ευχαριστώ. Για τους μετρήσιμους στόχους βεβαίως ε, μετρήσιμη στόχη μπορεί να είναι η αύξηση των προστατευόμενων περιοχών ωκεανών και θαλασσίων λεκανών κατά 30% ας πούμε, αλλά νομίζω ότι οπωσδήποτε εδώ πέρα θα είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά τους ε, στόχους της βιοποικιλότητας του 2030 να τους συζητήσουμε και με την Επιτροπή, πώς τα βλέπει η Επιτροπή ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε εφαρμογή όταν μιλάμε για δεσμευτικά νομικά μέτρα. Υπάρχουν πολλά τέτοια τα οποία δεν εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Και η μηδενική ανοχή για την μη ε, εφαρμογή. Ε, αυτό πρέπει να γίνει. Για τους στόχους θα υπάρξει μια στρατηγική βιοπικιλότητα, αλλά βεβαίω ε, δεν την έχουμε ακόμα. Είμαι ανοιχτό ε, να την ε, συζητήσω με την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νίκλας Χέρπστ για το ΕΛΚ. Θα ήθελα να εστιάσω, εδώ είμαι, στη δική μας ε, την περιοχή. Έχουμε κρίση στην περιοχή. Ε, δεν προκαλείται από την αλήθεια όμως. Και τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να πάρουμε για την ε, Βαλτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουν υπεραπορροφηθεί πόροι και δεν μπορούμε να στήσουμε παραπάνω και αν δούμε τις προτάσεις Υπάρχουν εταιρείε και αλήσα και από τη Δανία και από τη δική σας τη χώρα, τη Βαλτική, τις χώρες Βαλτικής, την Πολωνία, ε, άνθρωποι οι οποίοι θα πέσουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν φταίνε σε τίποτα. μπορεί να υπάρξει αλλαγή δραστηριότητα, ίσω ε, πώ μπορούν γρήγορα και χωρί γραφειοκρατία να διορθωθούν τα προβλήματα. Και δεν μιλάω για το πολιετέ το επόμενο, Εκεί καλά πάνε τα πράγματα. Εγώ μιλάω για του χρόνου όμως. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτού τους ανθρώπους που χωρί να, το, να φταίνει σε τίποτα θα μπουν σε τόσες δυσκολίες. Thank for... Σας ευχαριστώ. Πράγματι, αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα προβλήματα, εφόσον βέβαια εγκριθώ στη θέση του Επιτρόπου, που θα πρέπει να αντιμετωπίσω. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ήδη έχει ξεκινήσει διάλογο με τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Μήπως μπορούμε να βρούμε δηλαδή κάποιους πόρους για να παράσχουμε οικονομική υποστήριξη στους ε, ανθρώπους αυτούς. Τελειώνει βέβαια η τρέχουσα περίοδος ε, και δύσκολο θα είναι. Ε, θα αγωνιστούμε για να κινητοποιήσουμε ό,τι διαθέσιμους πόρους υπάρχουν. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα βρεθεί λύση από την ε, μέχρι τώρα Επιτροπή. Αν εγώ επιβεβαιωθώ, θα συνεχίσουμε το διάλογο για να δούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις που μπορούμε να ε, βρούμε. Δεν είναι εύκολο το θέμα και πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση αλλά δεν μπορεί να λήξει ε, η προσπάθειά μας φέτος. Δεν είναι μόνο για φέτος το, πρόγρα το πρόβλημα. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον ε, γάδο, τον ε, ανατολικό κυρίως και άλλα αποθέματα τα οποία φθήνουν και τι πρόβλημα υπάρχει για αυτούς τους αλείς που δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι και οι κοινότητες, οι παράκτες θα πληγούν πρώτα από όλους ε, αυτούς επηρεάζουν οι αλλαγές πιο πολύ, τους πλέον ευπαθείς. Για αυτούς θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Μπορεί να μην είναι εύκολο αυτό. Υπάρχουν τα διάφορα εργαλεία της επανεκπαίδευσης, επιμόρφωσης για να βρουν άλλες ευκαιρίες σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Και δική σας περιοχή ε, έχει τουρισμό πολύ επίσης. Είναι μια διέξοδος ίσως. Να προσθέσω κάτι. Δεν είναι το πρόβλημα υπεραλήψη, αλλά είναι άλλοι οι λόγοι, όπω είναι αλλαγή του κλίματος, για παράδειγμα, για αυτή την κατάσταση πέφτει Θα υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στην Κομισιόν. Να μην... Περιοριστούμε σε ένα μόνο ε, εργαλείο. Πράγματι, λέει ο κύριο ε, Σινκεβίτσιους, η κλιματική αλλαγή είναι πίσω από αυτή την κατάσταση στη Βαλτική. Ε, έχει αυξηθεί θερμοκρασία και αυτό επηρεάζει τα αποθέματα του γάδου, ε, εξού και η βιομάζα όχι φτωχοί απλά είναι, ε, αλλά σχεδόν ε, θα εξαφανιστούν τα αποθέματα γάδου σύντομα. Πρέπει πράγματι να ακολουθήσουμε ολιστική προσέγγιση. Υπάρχουν εργαλεία, αλλά και η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στην Αλία. Οι γεωργικές δραστηριότητες, ας πούμε, έχουν και αυτές σημαντικό ρόλο. Τα φυτοφάρμακα, τα ζανιοκτώνα, τα λοιπάσματα επιδεινώνουν και αυτά την κατάσταση στη Βαλτική. Ευχαριστώ για την ομάδα Ρινιού η Μαρία Ροδρίγες Ράμο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, πράγματι αναλάβατε τη δρομολόγηση της νέας στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα. Κύριε Φοντελάιν, Μιλάει για νέα μέτρα βιοπικιλότητας στον τομέα της οικονομίας, της γεωργίας, της παραγωγής. Δύο σημαντικά προβλήματα έχουμε. Το ένα είναι ο προϋπολογισμός και εσείς το αναφέρατε, είναι όμως τεράστιο το ζήτημα, διότι είναι ανεπαρκέστατος ο προϋπολογισμός για την προστασία της βιοπικιλότητας. Στο δίκτυο Natura χρειάζονται 6 δις, αλλά μόνο το 20% καλύπτεται. Και δεν μιλάμε μόνο για την αύξηση του προϋπολογισμού, πρέπει να υπάρχει και αποτελεσματικότητα σε ενεργές μας. Η μη τήρηση, η μη σωστή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων των ευρωπαϊκών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα από τα κράτη-μέλη, κάθε χρόνο προκαλεί 55 δις κόστος λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης ναι. και προβλημάτων υγείας. Εσείς θα θεσμευτείτε στο πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στη στρατηγική βιοπικιλότητα ε, ε, θα περιληφθεί αύξηση του προϋπολογισμού και θα υπάρξουν μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου παρακολούθηση και εφαρμογή τη κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Γιατί η Κομισιόν είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και του κοινοτικού κεκτημένου. Αυτή πρέπει να φροντίσει γι' αυτό απάντησα. Σε ευχαριστώ. Σε ό,τι τον προπολογισμό, βεβαίως και θα ζητήσω στεναρά και μετεπιτάσεως αύξηση του προπολογισμού. Θα συνεργαστούμε με τον Αντιπρόεδρο Φραν Τίμερμαν και με άλλους επιτρόπους. Και η ίδια η κυρία Βαντρελάιν νομίζω πολύ ξεκάθαρα δήλωσε ότι είναι στρατηγικό στόχος στρατηγικοί στόχοι πρέπει να έχουν και πάρει χρηματοδότηση, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι. Φυσικά την απόφαση δεν πάρει το σώμα των επιτρόπων συλλογικά και θα έχουμε συνομιλίε, διαβουλεύσει για να δούμε πού θα είναι προτεραιότητε, Η βιοπικιλότητα όμω. αν δείτε τις βασικές προτεραιότητες, η βιώσιμη ανάπτυξη, οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, είναι το κλειδί. Αν μιλάμε για την ε, κλιματική αλλαγή. έκθεση του ΕΑΗ λέει ότι η βιοπικιλότητα αν δεν διατηρηθεί θα ε, είναι υπεύθυνη για το 37% της κλιματικής αλλαγής. Άρα, σίγουρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και αν δεν αναλάβουμε, θα μας κοστίσει πολύ περισσότερο. Περιβαλλοντικές απώλειες, ε, η κυρία Φοντελάιν τα είπε ξεκάθαρα, το λέει και στην επιστολή ανάληψης ε, καθηκόντων. Μηδενική ανοχή για μη συμμόρφωση. Αυτό είναι σημαντικό. Και το έχω πει. Το είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Θα εξετάσω το σύνολο τη εργαλειοθήκη μας. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του διαλόγου, αυτό είναι το πρώτο. Αλλά αν δεν μας μείνει κάτι άλλο και αν δεν επαρκούν τα άλλα μέτρα, θα εξετάσουμε και το ενδεχόμενο της διαδικασίας επί παραβάση, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Sí. Por eh, Τέλος στη διάρκεια της δικής σας θητείας θα μπορούσαμε να περιμένουμε ένα νέο φιλόδοξο εργαλείο, μηχανισμό για την προστασία των δάσων, όχι των ευρωπαϊκών, μόνο, ε, των ευρωπαϊκών δασών, αλλά των δασών και χωρών που πλήττονται από τη δική μας την κατανάλωση. Έχετε προβλέψει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για τη βελτίωση της πιστοποίησης των λυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού ε, προϊόντων ε, που δεν θα είναι προϊόν αποψήλωσης των δασών. Απάντηση σε ό,τι αφορά την απορρίμωση των δασών, την ε, υποψήλωση των δασών. Φυσικά και πρέπει να δούμε τι αποτύπωμα αφήνουμε και θα συνεργαστώ με τους άλλους επιτρόπους, γιατί είναι σημαντικό. Η χρηματοδότηση, οι πόροι που δίδονται σε άλλες χώρες, να μην είναι τελικό δίκαιο στην αποδάσωση. Και το δεύτερο, πρέπει να βελτιώσουμε την επισήμανση. Θέλουμε αλυσίδες εφοδιασμού χωρίς αποψήλωση δασών. Και φυσικά εγώ θα αργωνιστώ γι' αυτό. Thank you ευχαριστούμε. Σίντζιτς. Um, Vi, ε, gospodine Sinkevičius, dolazite iz Litve. Κύριε προέρχεστε από την Λιθουανία και είστε ο υποψήφιος ε, επίτροπος για το περιβάλλον και τους ωκεανούς και Έχω να θέσω μια ερώτηση που δεν έθεσε άλλο συνάδελφο. Τι γίνεται όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με αυτού που ασχολούνται με ακτινοβολία. Με την ακτινοβολία. Ποιο συγκεκριμένο, είναι θέμα αυτό στην ε, Κροατία. Από το 1998, πάνω από 20 χρόνια υπάρχει θέμα τέτοιο στην Κροατία. Έχουμε μια διεθνή επιτροπή που ασχολείται με αυτό το ζήτημα, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα θερμικής ενεργείας. Όμως, η έρευνα που έγινε στο μεταξύ απεκάλυψε και άλλα ζητήματα και άλλους παράγοντες, ε, ιονίζοντες, ε, μη θερ, θερμικούς τέλος πάντων. Επίσης αυτό έχει να κάνει και με τους διαταράκτες ε, και έχουμε τελικά μια συνέργεια όλων των παραγόντων και είναι το αποτέλεσμα σορευτικό. Τι γίνεται, έχουμε νέες τεχνολογίες. Οπότε το πρόβλημα παροξύνεται. Θα λάβετε υπόψη αυτή την 20 ετία επιστημονικών διαπιστώσεων και να κάνετε κάτι για καλύτερη προστασία όσον αφορά την ακτινοβολία. Σας ευχαριστώ. Μη θερμική ακτινοβολία λέτε. Ε, βέβαια, δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά και ο ήλιος ε, δίνει μια τέτοια ακτινοβολία, εκπέμπει μια τέτοια ακτινοβολία και διάφορες... Ε, ε, ανθρώπινες δραστηριότητες, οι διαταράκτες, 3G, ε, 4G κλπ. Και έχουμε τάξει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Είπαμε επίσης για την φιλοδοξία της μηδενικής ρήπανσης. Επίσης και τα φυτοφάρμακα πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό και ενισχύουμε οικονομικά την βιολογική γεωργία. ένα και περισσότερο, βεβαίω και είμαι πρόθυμο να ακούσω του επιστήμονε, πάντα είμαι πρόθυμο να μελετήσω τι λένε και έχουμε τον ΠΟΗ, ο οποίο ε, είναι ενημερωμένο, παρακολουθεί τέτοια ζητήματα μονίμω και έχουμε τι συμβουλές που παρέχονται προ τα κρατημέλη για τέτοια ζητήματα. Και αν τελικά να λάβω αυτό το χαρτοφυλάκιο, βεβαίω και θα ακούω τι λένε οι επιστήμονες για τέτοιες απειλές που αφορούν ε, την ανθρώπινη υγεία. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι θέλετε να πάτε σε όλη την Ευρώπη και εγώ σας καλώ στην Κροατία όπου δυστυχώς Έχουμε κάθε μέρα άλλο ένα και περισσότερε κεραίε κινητών. Οι αρχέ δεν κάνουν τίποτα. Είναι το μόνο κράτο που δεν χρειάζεται άδεια για να στήσει κανεί κεραία κινητή τηλεφωνία. Και στο Ζάγκρεπ έγιναν κάποια απογραφτικά μέτρα για κάποιες παράνομες εγκαταστάσεις από το Σεπτέμβριο του 2008 υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Είπαμε να μην υπάρχουν κεραίες κοντά σε νοσοκομεία, σε σχολή. αλλά δεν τηρούνται όλα αυτά. Εδώ και 10 χρόνια το Υπουργείο Υγεία θα έπρεπε να έχει καταγράψει αυτέ τι κεραίε και να φροντίζει για την προστασία, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα ο Επίτροπο. Σα ευχαριστώ. Πήγα στην Κροατία πριν από δύο χρόνια πήγαμε τη σύζυγο. Ένιωσα το πόσο φιλόξενοι είστε. Ε, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μελέτη επιπτώσεων. Αυτό προβλέπεται από την ομοθεσία όλων των κρατών. Βέβαια υπάρχουν ε, κάποια περιθώρια, κάποια ευελιξία, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι κενό για να δημιουργούνται προβλήματα εις βάρος της υγείας. Thank you. Ε, for SND, Mohamed... Και τώρα, Μοχάμεντ Σαχίμ για τους σοσιαλιστές. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε υποψήφιοι επιτροπή, οι μελέτες έχουν δείξει ότι μια στρατηγική κυκλικής οικονομίας μπορεί να μειώσει τις ε, εκπομπές Ευρωπαϊκής Ένωσης του μισό. Κατά την τελευταία θητεία το Κοινοβούλιο και οι σοσιαλδημοκράτες σας πίεσαν για να, βάλετε, για να δημιουργήσετε πολιτικές προς μια κυκλική οικονομία. Όμως οι δράσεις εστίασαν περισσότερο στην φάση του τέλους κύκλου ζωής, ενώ πρέπει να δείτε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, από τον σχεδιασμό. Ήδη έχοντας αυτό κατά νου, πώς σκοπεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στο να επιτύχει μια μη τοξική κυκλική οικονομία. Θα, σχε... θα νομοθετήσετε εκ νέου ή θα διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ε, της υφτάμενης ε, οδηγίας επιπλέον οι νέοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για το ότι πετάμε τα καταναλωτικά προϊόντα, ειδικά τα ρούχα. Τι προτείνεται στο πλαίσιο της κυκλικής ε, οικονομίας ε, σε σχέση με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Η κυκλική οικονομία είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει βιωσιμότητα και το βασικότερο για να ξαναχρησιμοποιούμε τους σπόρους μας. 88% των πόρων μας α, πετιούνται. Μόλις 12% ξαναχρησιμοποιούνται, οπότε έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Και πρώτα απ' όλα βεβαίως πρέπει να δούμε όλες τις φάσεις αυτού του κύκλου, από τον σχεδιασμό, γιατί συνήθως, σωστά είπατε, ότι ήδη από τη φάση του σχεδιασμού η συσκευή ή το οτιδήποτε σχεδιάζεται για να κρατήσει λίγο και να πεταχτεί. Και έτσι δεν μπορούμε να το αποσυναρμολογήσουμε και να αλλάξουμε μπαταρία ή οθόνη ή μικρόφωνο. Οπότε πρέπει να δούμε το θέμα στη φάση του σχεδιασμού. Και εδώ πέρα ακριβώς ε, ο καλύτερο τρόπο να γίνει αυτό είναι να αλλάξουμε τον σχεδιασμό, να έχουμε μεγαλύτερου κύκλου, αλλά πρέπει να δούμε και τι μικρομεσαίες επιχείρησει. Έχω ένα πολύ καλό παράδειγμα που ίσω το ξέρετε. Ε, υπάρχει μια εταιρεία στη Λιθουανία, Winted, που ξεκίνησε μια πλατφόρμα για να πουλάει ρούχα βασικά. Κάτι το οποίο έχει τεράστιε δυνατότητε. Βλέπω χρησιμοποιείται σε Βέλγιο, Γαλλία και σε άλλε χώρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κυκλική οικονομία να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες. Ψηφιοποίηση λοιπόν είναι μια ευκαιρία. Το blockchain. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τους πόρους, ε, τα υλικά, να υπάρχει ένας πραγματικός κύκλος. Επίσης ο τομέας των κατασκευών που είναι υπεύθυνο για το 1 τρίτο ε, των αποβλήτων. Και αυτό θα είναι προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης. Σας ευχαριστώ. Έχω και άλλη μια ερώτηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να σταματήσει η ρήπανση από τα πλαστικά. Τι σκοπεύετε να κάνετε, όχι μόνο για τα μικροπλαστικά που ε, πετάγονται εσκεμένα και βρίσκονται μεταξύ άλλων στα καλλιτικά, αλλά και στα μικροπλαστικά που παράγονται μη ηθελημένα. Στη γραπτή σας απάντηση μιλάτε για ε, τις πράσινες δημόσιες προμήθειες. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουμε ότι οι βιώσιμες ε, δημόσιες προμήθειες ε, περιλαμβάνουν και την κοινωνική διάσταση. Μπορούμε έτσι να ε, περάσουμε στην κυκλική οικονομία. Ποια μέτρα θα λάβετε για να περάσουμε στις βιώσιμες δημόσιες προμήθειες. Ως υπουργός ε, εγώ ενεθάρρυνα τι ε, καινοτόμε ε, δημόσιε προμήθειε. Ήμουν υπεύθυνο ε, για τις δημόσιε προμήθειες και πραγματικά αισθάνεται τελείω διαφορετικά ο κόσμος. Πρέπει νομίζω να μετακινηθούμε. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν στόχου, δηλαδή πόσο τη 100 θα έχουμε πράσινε προμήθειε. Βεβαίω μπορούμε να βοηθήσουμε και εμεί. Όσον αφορά τώρα τα πλαστικά, όπως είπα, ε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε το ότι ε, φτιάχνετε κάτι σε 5 δευτερόλεπτα, το πετάμε σε 5 λεπτά και κάνει 500 χρόνια να διαλυθεί. Ε, βιοδιασπόμενα, μικροπλαστικά και βεβαίως να μην είναι τοξικά για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά στην κυκλική οικονομία. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, Δύο ώρες μιλάτε. Ε, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Έχουμε τις τελευταίες πέντε ερωτήσεις. Πλησιάζουμε στη γραμμή του τερματισμού. Κυρία Τότ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος όσον αφορά την προστασία της ε, βιοπικιλότητας. Όμως δεν επαρκεί αν το κάνει μία ήπειρος μόνο. Θεωρώ ότι χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία. Η αποστολή σας θα είναι να συνεισφέρετε του χρόνου στην ε, Κίνα να εγκριθεί μια φιλόδοξη συμφωνία και μια πρόταση για την βιοπικιλότητα μέχρι το 2030. Στις ε, γραπτές σας απαντήσεις βλέπουμε πώς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στην διεθνή σκηνή, στον αγώνα κατά της μείωσης της βιοπικιλότητας. Πώς θέλετε να το επιτύχετε αυτό, έχετε συγκεκριμένα σχέδια. Πώς θα παρακινήσετε τις τρίτες χώρες να προστατεύσουν ε, ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Βεβαίως, είναι σημαντικό να έχουμε φιλόδοξους στόχους και για να έρθουν και άλλες χώρες με το μέρος μας ε, πρέπει να ηγηθούμε δια του παραδείγματος. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική φιλοδοξία η οποία όμως θα εφαρμόζεται κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, βεβαίως, είναι σημαντικό να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Είναι δύσκολο να πούμε τώρα ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι στόχοι. Πρέπει να έχουμε διάλογο με τους εταίρους μας, με τις χώρες. Οπωσδήποτε θα αναζητήσω σύμβουλες και εάν με ορίσετε θα πάω στην Κινά, δεν θα είμαι μόνος μου. Με μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας για να έχουμε μια ισχυρή θέση και βεβαίως μια συζήτηση και ένας διάλογος για τους πιθανούς στόχους. Όταν ε, το σκεπτόμουν ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι στόχοι, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι καλό στόχος θα ήταν να έχουμε ένα 30% προστατευμένων περιοχών στον κόσμο και επιπλέον ε, να έχουμε ένα ξεχωριστό άρθρο ε, για την Αρκτική ε, βλέπουμε ότι οι αλλαγές στην Αρκτική με τον πάγο που λιώνει σημαίνει ότι ασκείται περισσότερη πίεση στην περιοχή αυτή του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει βιωσιμότητα και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Έτσι ε, βλέπω εγώ, την φιλοδοξία που θα πρέπει να έχω στην ε, Κίνα. Βεβαίω, ε, όπω είπατε, θα είμαι στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε, αλλά είναι σημαντικό και οι εταίροι μας να ακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρατε και το ότι είναι σημαντικό σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης να αντιμετωπίσουμε την υποβάθμιση της ε, βιοπικιλότητας. Ε, Και αναφέρατε ένα παράδειγμα στις ε, γραπτές σας απαντήσεις Μιλήσατε για τις διεθνείς εμπορικές ε, συμφωνίες ε, ε, και ότι πρέπει να περιλαμβάνουν αυστηρότατες περιβαλλοντικές ρήτρες. Τα κράτη-μέλη, τα τρίτα όμως, πώς μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε ότι θα εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους και τι θα κάνετε αν ένα τρίτο κράτος δεν τήρει τις δεσμεύσεις του. Thank you. Uh, first of all, of course, it is, it's going to be Πρώτα πρώτα είναι σημαντικό να συνεργαστούμε στενά με τον Φιλ Χόγκαν, τον Επίτροπο για τα εμπορικά θέματα και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα θέσουμε και στον ΠΟΕ. Ε, βέβαια, η βιωσιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι που έχουν προσυπογράψει 197 χώρες να είναι κοινό στόχο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά ενός με τον Επίτροπο Εμπορίου. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι χρειάζεται και να προστατεύσουμε και την αγορά. και να δούμε πού η προσφορά δεν είναι βιώσιμη. Κύριε Κόρμπετ, για το σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε για τους ωκεανούς. Εγώ θα προσέθετα και τις θάλασσες. Για βάλτε το γι' αυτό στον τίτλο του χαρτοφυλακή. Δεν θα συμφωνούσατε ότι η ρήπανση από απορρίμματα των θάλασσών είναι η μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον και επίσης ε, βράβει πάρα πολύ ε, τις ε, κοινότητες των παραλίων. Όλα αυτά καταλήγουν στα δίχτυα των αλλιών συνήθως. Θα πρέπει να πληρώσουν για να διατεθούν αυτά τα απορρίμματα και αυτό σιγά σιγά αλλάζει και το IMFF επίσης είναι υπέρ του να γίνουν επενδύσεις ούτως ώστε να καθαριζονται οι θάλασσες και υπάρχει μια κάποια επιτυχία περιορισμένη από αυτά τα μέτρα. Μήπως τώρα χρειάζεται όμως να υπάρξει κάποιο είδους ε, σφαιρικότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, για το, την διάθεση και καταστροφή αυτών των απορριμμάτων από τη θάλασσα. Εσείς αυτό το πρόβλημα πώς θα το αντιμετωπίσετε, Επίτροπος. Είναι σημαντικό σύμφωνα με το Green Deal κατά την θητεία μου να κάνω την μπορώ τόσο ώστε να είναι καθαρές, ε, να είναι υγιείς και βιώσιμες οι θάλασσες αλλά και οι ωκεανοί. Πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του 30% για το Natura 2000 ε, και βέβαια και πέρα από το 30% των προστατευμένων περιοχών θα πρέπει να υπάρχει προστασία, να υπάρχει σωστή εφαρμογή των όσων προβλέπουμε και αυτό δεν σημαίνει ότι αν μια περιοχή προστατεύεται από τον 2000 δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κάποιες οικονομικές δραστηριότητες όπως ε, η αλία, κάθε άλλο. Ε, βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουμε τη βιώσιμη αλία και σε σχέση με τη μείωση της ε, ε, ρήπανσης, ε, τότε θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και να μην διασπαθίζουμε πόρους που αξίζουν. Θα πρέπει να τους στρατεύουμε για, τους για την οικονομία μας. Τώρα όσον αφορά τα κίνητρα προς αλλιείς, αυτό γίνεται από πολλές χώρες, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. θα πρέπει όλες τις δραστηριότητες τους να είναι βιώσιμες, ό,τι χρειάζεται να καθαρίζεται κλπ. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με, με διάλογο και έτσι να δοθούν κίνητρα για τους βιώσιμους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. This and many of the other issues addressed Ίσως χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει και άλλα μέτρα. Πάντως, στην επιστολή σας λέτε ότι θα κινηθείτε επί τη βάση του ότι θέσπιση μέτρου σημαίνει την κατάργηση προϋπάρξαντος ανεξαρτήτω του τιμήματο των επιπτώσεων. Και εσεί τι λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει κάθε μέτρο να αξιολογείται όχι από τη βάση ε, κάποιων ε, πιστεύω στατιστικών, αλλά επί τη βάση της ουσίας του μέτρου. Επίτροπο, σας ευχαριστώ για αυτό που ερωτήσατε. Ως Υπουργός Οικονομικών και Καινοτομίας είχα ασχοληθεί πολύ για να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αλλά δεν μπορεί να είναι μηχανιστική η διαχείριση του θέματος. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, όπως το είπαν και οι άλλοι υποψηφοί επίτροποι και θα σιγουρέψω το ότι θα καταπολεμήσω την γραφειοκρατία χωρίς να απονευρώσω την περιβαλλοντική μας νομοθεσία. και για τη βιοπικιλότητα και γενικά έχουμε φιλόδοξους στόχους και οι οποίοι θα επιβλεχθούν μόνο εάν η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους. The very much. Thank you very much for your answers. Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε μέχρι τώρα και μας είπατε ότι θα κινηθείτε και προς την κυκλική οικονομία και προς ε, πιο καθαρές θάλασσε, άρα θα έχετε μέθοδο την συνέργεια. Σύμφωνα με το 7ο πρόγραμμα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποια υλικά μη τοξικά και αυτά να είναι ανακυκλώσιμα και να είναι πηγή πρώτων υλών. Δυστυχώ, η προηγούμενη ε, Κομισιόν έκανε το αντίθετο. Αδειοδότησε κάποια πολύ, τοξικά, ε, πολύ που δεν ήταν και ανακυκλώσιμα αυτό στρέφεται κατά του περιβάλλοντος, γιατί αυτά τα τοξικά υλικά μένουν πάρα πολύ χρόνο γύρω μας. Και τι θα γίνει με τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών. Δηλαδή θα κάνετε κάτι ταυτόχρονα με την κυκλική οικονομία και ε, ε, την ε, ρήπανση δηλαδή να αντιμετωπίσετε με την κυκλική οικονομία ε, αυτές τις βλαπτικές ουσίες και να τις κάνετε ανακυκλώσιμες. Ο Επίτροπος, ευχαριστώ. Υπάρχει σαφής σχέση με το σύλλο του χαρτοφυλακίου και αυτά που λέω στην Επιτροπή, δηλαδή τη μηδενική ε, μόλυνση, βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία, ε, όλα όλα αυτά μέσα στο χαρτοφυλάκιο υπάρχουν και αν ένα από αυτά το βγάλουμε δεν θα προχωρήσουν τα υπόλοιπα στοιχεία. Άρα όλα αυτά θα είναι ο κεντρικός άξονας στο New Green Deal. Η μηδενική μόλυνση φυσικά και συνδέεται με μια στρατηγική κατά των τοξικών υλικών και ουσιών. Μόνο αν δεν διασπαθήσουμε τους πόρους μπορούμε να τους ξαναχρησιμοποιήσουμε και να τους ανακυκλώσουμε. Επίσης, η κυκλική οικονομία θα πετύχει μόνο άπαξ και βρούμε έναν τρόπο να έχουμε έναν κύκλο χωρίς τοξικά. Επομένως, τα πλαστικά τα οποία προέρχονται από φιλικές, ας τις πούμε, χημικές ουσίες και να ξέρουμε ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους και να χρησιμεύουν για μια σειρά σκοπών. Να, πώς μπορεί να αποδώσει η κυκλική οικονομία. Και βέβαια και εγώ θα κινηθώ προς τα εκεί. Thank you. Uh, uh, the European Parliament has objected... Έξι φορές μέχρι τώρα είχαμε ένσταση για κάποιες αδειοδοτήσεις της Κομισιόν. Και στην Σουηδία η κυβέρνησή μας, στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, επίσης πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε την υπόθεση κατά της Επιτροπής για ε, κάποιες αδειοδοτήσεις που εκρήθησαν παράνομες. Και σας ρωτώ, εσείς, τι θα κάνετε στη συνέχεια εκείνων των ενστάσεων μας, θα κάνετε κάποια αλλαγή ε, πορείας, ε, που θα λάβετε υπόψη αυτές τις αποφάσεις και όσον αφορά το REACH θα εφαρμόσετε αυτά που προβλέπονται για αυτά τα υλικά. Το REACH είναι μια πάρα πολύ βασική νομοθεσία. Καλύτερη στον κόσμο για αυτούς τους σκοπούς. Ε, βέβαια θα συμμορφωθούμε όλα αυτά έχουν γίνει και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτά τα μέτωπα που είπατε, όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ περιμένω πώς και πώς. Το ΡΙΤΣ να καλύψει και αυτό τον βασικό άξονα Έχουμε τη στρατηγική κατά των τοξικών και των χημικών. Και όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, όλα αυτά τώρα είναι υπομελέτη. Μόλις ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας θα προχωρήσουμε. Bilbao for Renew Europe. Πρόεδρε και κύριε υποψήφιοι επίτροπε, Οι γυναίκε που ασχολούνται με την αλληλεία θέλουν τη βοήθειά σα και οπότε θέλουμε και αυτέ να τις καλύψετε στο χαρτοφυλακείο σα και με το χαρτοφυλακείο σα. Εμεί συνεχίζουμε τον κανονισμό για τον έλεγχο και θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα για το πρώτο κομμάτι αυτή τη θητεία και εσεί αναφέρατε στην εισήγησή σα ότι χρειαζόμαστε αυστηρού κανόνε για τα αλληλευτικά προϊόντα και μα είπατε και για το δίκτυο το και το δίκτυο. Και για αυτό το για τη διαδρομή του προϊόντος από το δίχτυ στην κονσέρβα. Έχουμε επομένω μια σειρά προϊόντων τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλή ποιότητα, οπότε έχουμε την ανιχνευσιμότητα στις ετικέτες των ε, κονσερβών και θα πρέπει όλα αυτά στην ε, αξιακή αλυσίδα να αναβαθμιστούν και να εξασφαλιστεί ε, εισόδημα για τις κοινότητες των αλλήλων. Και οι καταναλωτές επίσης θα πρέπει να ξέρουμε από την ετικέτα τι αγοράζουμε και τι καταναλώνουμε εσείς. Πώς το βλέπετε. Θα κατεβάσετε κάποια νομοθετική πρόταση ούτως ώστε να τα καλύψετε όλα αυτά. Νομίζετε ότι η περιφερειοποίηση των αλληλευτικών ταμείων μπορεί να βοηθήσει τον ρόλο ανδρών και γυναικών της παράκτειας αλληλείας και επίσης να είναι επικερδής δραστηριότητά και νομίζετε ότι θα προστατεύσετε αυτήν την περιφερειοποίηση. Και σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος. Πρώτα, απ' όλα για τις γυναίκες και το ρόλο τους. Σε μια έκθεση πρόσφατα φάνηκε πόσο σημαντικό είναι και θα συνεργαστούμε με τον Αρμόδιο είναι ένας τομέας που πρέπει να γίνει ελκυστικός για όλους, να υπάρχει επίσης σεβασμός για όλους. Η μεταποίηση επίσης ε, είναι πολύ σκληρή δουλειά και δεν αμείβεται όσο ε, το ψάρεμα πάντοτε. Άρα και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Στο ό,τι αφορά την χλασιμότητα, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε ποιοτικό, ποιοτικά τρόφιμα, καλά τρόφιμα και πρέπει τα υψηλά μας πρότυπα να διατηρηθούν. Και η επισήμανση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρει ο καταναλωτής δηλαδή τι αγοράζει. Η πράσινη ετικέτα κάτι να σημαίνει και η χνησιμότητα είναι σημαντική. Από το δίχτυ, όπως είπα, μέχρι την κονσέρβα. Έχουμε και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, την ψηφιοποίηση, τα ψηφιοποιημένα εργαλεία. Να βοηθήσουμε τους εταίρους μας επίσης να χρησιμοποιήσουν προγράμματα όπως το ΚΑΤΣ και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να έχουμε συνομιλίε που θα οδηγήσουν σε καλύτερα πρότυπα αγορά και σε καλύτερη επισήμανση. Τα δικά μας πρότυπα σίγουρα είναι ψηλά και πρέπει να τα διατηρήσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Πράγματι είναι σημαντικό οι γυναίκες να την υπόψη και για την ένταξή τους θα πρέπει να αναγνωρίζονται και επαγγελματικέ γνώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αναφέρεται αυτό, ούτε αυτή την κλασιμότητα. Πράγματι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Εσείς όμως δεν θέλω να μου λέτε μόνο αν θα προχωρήσετε και θα δουλέψετε από αυτού, αλλά αν συμφωνείτε ότι η προέλευση των προϊόντων πρέπει να μπει στην ετικέτα. Αυτό ζητάμε. Και το δεύτερο για την περιφερειοποίηση των ταμείων, των κονδυλίων. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση και θα ανταποκριθεί και στο να έχουμε συνεκτικούς στόχους στην αλληλευτική πολιτική. Απάντηση. Η προέλευση πράγματι, όπως είπατε, είναι σημαντική. Όμως, πρώτα απ' όλα, αυτά που γράφονται στην ετικέτα πρέπει να είναι πραγματικές πληροφορίες, αληθείς πληροφορίες. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης για την αγορά μπορεί να το πετύχουμε αυτό. Αλλά πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ακριβώ την περιέχει το προϊόν και μετά να το περιλάβουμε στην ετικέτα για να μπορεί να κάνει τεκμηρωμένες επιλογέ ο καταναλωτή. Περιφερειοποίηση. Το είπα και πριν. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Και χρησιμοποιείται ήδη πολύ για τη λεκάνη της Μεσογείου τώρα και θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Θέλουμε την ε, στήριξη των γνωμοδοτικών συμβουλίων και αυτό διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων κρατών που μοιράζονται την ίδια Και σιγά σιγά φτάσαμε στην παρελθόν 25 ερώτηση και τον κύριο Βαντάλεν. Προσδεθείτε. I will turn to Dutch. Τώρα θα μιλήσω Ολλανδικά. Voorzitter, ehm, dit parlement en το Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή Αλίας ε, διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας η Κομισιόν είναι κατά της θέσης του Κοινοβουλίου γιατί φοβάται ότι η θέση μας θα οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι δυσάρεστη για τα αποθέματα. Στην ε, χώρα μου λοιπόν Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί νέα καΐκια ε, τα οποία είναι και υβριδικά συν της άλλης ε, λοιπόν δεν υπάρχει φόβος με αυτά τα καΐκια για υπεραλίευση γιατί τηρούν τα πάντα και τις ποσοστός και όλα. Λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξής το συγκεκριμένο. Γιατί φοβάστε τα νέα σκάφη τα οποία είναι καλά και για το περιβάλλον και για την αλληλεία. Ενώ θα έπρεπε να λέμε είναι καλά για το περιβάλλον, δεν εκπέμπουν καθόλου, προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Okay, uh, I understand, uh... Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα αφορούσε... Μιλάτε για την παράκτη αλία. Μιλήσατε για νέα σκάφη, ότι φοβόμαστε τα νέα σκάφη. Αν μπορείτε να το επαναλάβετε. Εγώ μίλησα για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για νέες ναυπηγήσεις. Τα, για νέα πλοία τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και είναι πιο επιλεκτικά στην αλία, αλλά είναι ακριβά. Και εμείς λέμε να χρησιμοποιηθεί το νέο Ταμείο Αλίας. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Για την χρηματοδότηση από το Ταμείο χρειαζόμαστε περαιτέρω συζήτηση γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να ξοδεύουμε το δημόσιο χρήμα. Είναι μια επένδυση που θα μπορούσε να έρθει από τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοί σας πριν ε, ζήτησαν για βελτίωση των ε, συνθήκων κάποια σκάφη είναι και 30 ετών, είναι και ζήτημα ασφαλεία. Είναι σημαντικό το θέμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η ναυπήγηση νέων σκαφών ε, συμβάζεται με τους ε, στόχους μας, ε, όπως έχουμε συμφωνήσει στην, στο Αλληλευτικό Ταμείο. Όσον αφορά τα πιο επιλεκτικά αλληλευτικά εργαλεία, πρέπει να το δούμε μέσω της έρευνας της επιστήμης, αλλά η βελτίωση. Και οπωσδήποτε εδώ πέρα μπορούμε να ε, επενδύσουμε δημόσιο χρήμα στην έρευνα για να μπορούν να ψαρεύουν οι ψαράδες μας πιο επιλεκτικά με τρόπο πιο βιώσιμο και να έχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, χρειαζόμαστε πλοία τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς εκπομπές και για μένα είναι σαφές ότι θα πρέπει να τα στηρίξουμε από το νέο Ταμείο Αλίες και ζητώ από εσά να μην έχετε ε, αυστηρή θέση ως Κομισιόν αλλά να στηρίξετε τον κλάδο να έχουμε καλά ε, σκάφη τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. And I agree with you. Ναι, συμφωνώ μαζί σας κύριε Φαντάλεν. Ε, πράγματι, ο στόχος είναι να έχουμε αποφάσεις φυσικές προς το περιβάλλον. Ως Υπουργός Οικονομίας μπορώ να σας πω ότι ε, οι μικρές επιχειρήσεις ε, θέλουν ε, χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη. Εκεί πέρα θα μπορούσε να ξοδευτεί δημόσιο χρήμα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Να τους βοηθήσουμε με την έρευνα, με τις αποφάσεις που μπορεί αργότερα να εφαρμοστούν. Δεν είμαι σίγουρος ότι... Εντάξει, η πρόθεση είναι καλή, αλλά δεν ξέρω αν θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Thank you all. Thanks all. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Ο υποψήφιος επίτροπος τώρα έχει την δυνατότητα να κάνει μια πεντάλεπτη δήλωση. Λοιπόν, έχετε, πλησιάζετε τη γραμμή του τερματισμού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε. Χάρηκα και για την δέσμευση που επιδεικνύετε και για τις ερωτήσεις που κάνετε. Βλέπω πως σας ενδιαφέρει το θέμα και σημειώνω πως η βιοπικιλότητα, η κυκλική οικονομία, οι ψαράδες, μικροί, μεγάλοι και οι σχετικές κοινότητες είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σας. Ελπίζω να ήμουν από την πλευρά μου σαφής για το ότι θέλω να συνεργαστούμε. Η βιωσιμότητα είναι κοινή μας ευθύνη. Η εντολή αυτή, η θητεία αυτή θα είναι η πιο πράσινη που έχει ποτέ η Ευρώπη. Αυτό το είδαμε από την προσέλευση στις ευρωεκλογές ε, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και από τις επιστολές που έστειλε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θα είναι γαλάζια η τελευταία έκθεση της ε, διακυβερνητική διάσκεψης για το κλίμα έδειξε πόσο σημαντική είναι η ωκεανή για το περιβάλλον μα. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο διατρέχει ολόκληρη την Κομισιόν ε, από το κλίμα και τους ωκεανούς μέχρι την αλληλεία, τη γεωργία, τις επενδύσεις, τι μεταφορές και την υγεία. Αλλά το θέμα δεν αφορά μόνο τι ε, πολιτικέ ή το περιβάλλον και οπωσδήποτε δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά το τι είδους κοινωνία θέλουμε. Αφορά τους ψαράδες που δεν μπορούν πλέον να βγουν να ψαρέψουν. Αυτούς οι οποίοι, τους οποίους έπληξε ο οικονομικός μετασχηματισμός. Θα ήθελα λοιπόν οι δικές μου πολιτικές να συνεισφέρουν σε μια πιο δίκαιη κοινωνία που δεν θα αφήνει κανέναν πολίτη πίσω. Θα ήθελα να διασφαλίσω ότι θα είμαστε επιτυχής, θα υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση. Χρειαζόμαστε στοχευμένα μέτρα για τους ευπαθείς. Θέλω να είμαι μέλος μιας ομάδας που θα πάει την Ευρώπη προς μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση, γιατί όταν είμαστε φιλόδοξοι δεν βελτιώνουμε μόνο το περιβάλλον, δημιουργούμε κοινωνική δικαιοσύνη. Βελτιώνουμε την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ζωή των πολιτών μας. όταν η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα για τη μόλυνση, δεν βλάπτει μόνο το περιβάλλον, βλάπτει την οικονομία, την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία των πολιτών μας. Σε πολλά μέτωπα λοιπόν έχουμε μια τεράστια ευκαιρία με το χαρτοφυλάκιο αυτό. Η πρόεδρος μας ζήτησε η Ευρώπη να είναι η πρώτη ήπειρος η οποία θα είναι κλιματικά ουδέτερη και ένας υγιής πλανήτης σημαίνει υγιές περιβάλλον και υγιείς θάλασσες. Τα θαλάσσια πάρκα προστατεύουν την βιοπικιλότητα, αλλά υπάρχουν και μακροπρόθεσμα ωφέλη για την αλληλεία. Και αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν οι ψαράδες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ωκεανούς μας αν δεν προστατεύσουμε και την ξηρά. Μια φιλοδοξία όπως η μηδενική ρήπανση θα επηρεάσει πάρα πολύ τι θάλασσε, Καθώ αυτά τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα ξεκινάνε από την ξηρά, η ρήπανση δηλαδή. Πάνω από το 40% των ειδών των θαλασσίων επηρεάζονται. Χρειάζονται βοήθεια, βιοπικιλότητα, μηδενική ρήπανση. Από το χωράφι στο πιάτο μα. Όλε αυτέ οι προτεραιότητε πρέπει να επιδιωχθούν από κοινού. Θέλω λοιπόν τη βοήθειά σα για να είμαστε πιο κοντά στου πολίτες, στις στο τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν τις δικές σας τις γνώσεις και την συμβολή σας όταν θα πηγαίνω στις ε, χώρες σας. Εσείς ξέρετε το τι γίνεται. Ο δασοπόνος ε, που προστατεύει τα δάση, οι ψαράδες που φοβούνται ότι θα εξαφανιστεί το αλίευμα. Εσείς είστε η γέφυρα με τους πολίτες ε, και ελπίζω να τα καταφέρω με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να πιείτε μια μπυρίτσα τώρα για να χαλαρώσετε κύριε Οριστέντα Επίτροπε. Και εμείς ε, και οι συντονιστές των δύο επιτροπών, ηρεμία, ησυχία, έλεγα λοιπόν ότι οι συντονιστές των δύο επιτροπών θα συναντηθούμε ε, καταρχάς στις 6 και στις 7 από κοινού για την αξιολόγηση.